Κυρίε και κύριοι, σα παρακαλώ να καθίσετε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά στην απογευματινή μας συνεδρίαση που λαμβάνει χώρα από κοινού με την Επιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με την Αντιπροσωπεία για τις ε, σχέσεις μας με τη Ρωσία. Χαίρομαι που βρίσκεται κοντά μας και ο πρόεδρος της Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας μάλλον, ο κύριος Ότμαρ Κάρας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κοντά μας τον κύριο Μίχαλ Κοντακόφσκι, ε, τον ιδρυτή του κινήματος Open Russia. Κύριε Κοντοκόφσκι, είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε στο Στρασβούργο, αλλά δεν έχουμε σαν τίποτε επίσημα. Νομίζω λοιπόν ότι για μας ε, είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να σας πούμε ότι την κατάχρηση δικαιοσύνης που έγινε στην περίπτωσή σας τη θεωρούμε απαράδεκτη. Το θεωρούμε απαράδεκτο ε, το ότι εκδίδονται τέτοιου είδους δικαστικές αποφάσεις ε, με τόσο μακρά διάρκεια κράτησης. Αυτό δεν εντάσσεται ε, σε ένα σύστημα δικαίου που να γνωρίζουμε εμείς. Και αυτή εξάλλου ήταν και η άποψη της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία σας χαρακτήρισε έγκλειστο για λόγους συνείδησης και από το 2013 μέχρι συγγνώμη, από το 3, 2003 μέχρι το 2013 ήσασταν σε έγκλειστο, σε φυλακή, σε καταναγκαστικά έργα. Μετά την απελευθέρωσή σας ε, βρήκατε το θάρρος να ε, αγωνιστείτε για την υπόθεση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία και μεταξύ άλλων με την ίδρυση του κινήματος Open Russia γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις ε, με τη Ρωσία και λόγω των πράξεών της στη γειτονική χώρα είναι σε κρίσιμο επίπεδο. Υπάρχουν και οι ε, στις κρίσεις στη Μολδαβία, στη Γεωργία και σε άλλες χώρες. Θα μπορούσα κάλλιστα να παριθμίσω πολλά, αλλά θα μας ενδιέφερε καταρχήν ιδιαίτερα να ακούσουμε τη δική σας την άποψη. Μας ενδιαφέρει μάλιστα ιδιαίτερα η δική σας η άποψη για το πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις ε, στο εσωτερικό της Ρωσίας, ε, πώς ε, κρίνετε το κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες δημοκρατικής συνεργασίας, ανοίγματο και γενικά κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών ε, κατά πόσο είναι δυνατόν να προχωρήσει αυτή η ε, διαδικασία ανεξαρτητοποίησης ε, των πολιτών στην Ρωσία. Κύριε Κοντοκόφσκι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι που με υποδέχεστε στην συνεδρίαση της Επιτροπής σας και θέλετε να με ακούσετε. Θα σας παρουσιάσω τις εντυπώσεις μου για τα τεκτενόμενα στην πατρίδα μου. Σήμερα το σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας αντιμετωπίζει τις πιο σημαντικές προκλήσεις μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως προς την ουσία, η ξεκάθαρη προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία και η λιγότερο σαφής ε, ε, προσάρτηση της ε, νοτιοανατολικής Ουκρανίας παραβιάζει τις συμφωνίες του Πότσδαμ. Και σίγουρα δεν είχαμε και μετά την Συμφωνία της Γιάλτας μεγάλη ηρεμία στην Ευρωπαϊκή. αλλά ούτε μία φορά α, κάποια από τα συμβαλόμενα μέρη της Γιάλτας δεν παραβίασε κατάφορα την κατάσταση τη μεταπολεμική με εμπόλεμες ενέργειες. Και τώρα θα πρέπει να δούμε αν όλα αυτά είναι σωστά και δίκαια ή όχι. Είναι θέμα αρχής. Οι ρωσικές αρχές για μία ακόμη φορά άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας και δημιούργησαν απειλές και κίνδυνο παρόμοιες με αυτές που έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο πολλές φορές. Και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτές οι εδαφικές βλέψεις ε, της Ρωσίας. Και μάλιστα μια ιστορία που ξεκίνησε στην Κρυμαία δεν είναι τυχαίο που τελειώνει στην Κρυμαία. Και αυτό που θέλει το Κρεμλίνο είναι να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση της ε, άνεσης που είχε, ώστε κανένας εξωτερικός παράγοντας να μην μπορεί να απειλεί, να υπονομεύει το καθεστώς. Και τα όρια και οι προοπτικές του καθεστώτος του Κρεμλίνου στρέφονται γύρω από τη συμφωνία του Ελσίνκη χωρίς όμως τρίτο πακέτο. Θέλουν ουσιαστικά να ανασκευάσουν όλη την ευρωπαϊκή ιστορία. Όχι από το τείχος, από τη βάση του τείχους του Βερολίνου, αλλά και 15 χρόνια πριν. Ουσιαστικά θέλουν να διορθώσουν την, ε, την ε, ευρωπαϊκή ιστορία. Και το Κρεμλίνο θέλει να επανέλθει στην πολιτική της ε, συνύπαρξης αποφεύγοντας οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις. Το κρεμίνο δηλαδή θέλει ε, να έχει το απόλυτο ελεύθερο στην ζώνη επιρροής του. Και από αυτή την άποψη το κρεμίνο δημιουργεί τεράστιες απειλές στην Ευρώπη γιατί έχει τεράστιο στρατιωτικό δυναμικό, έχει τέτοιο πλωστάσιο η Ρωσία που θα μπορούσε να καταστρέψει τον πλανήτη ορόκληρο. Και αν κάποιος το ξεχνάει, οι αρχές του Κρεμλίνου είναι έτοιμες να του το υπενθυμίσουν. Όλο αυτό το στρατιωτικό δυναμικό, το τεράστιο οπλοστάσιο που έχει η Ρωσία θα αναπτυχθεί και στο μέλλον. Και μάλιστα όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια ενός ανθρώπου που το η πνευματική του ικανότητα και το ηθικό του παράστημα βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Και η Ευρώπη θα πρέπει παρά την παράνομη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία να βρει μία μορφή διαλόγου γιατί οποιαδήποτε άλλη μη διπλωματική λύση μπορεί να οδηγήσει σε πολεμική σύραξη παγκοσμίων διαστάσεων. Όπως είπε βέβαια ένας σημαντικός Ρώσος στο του 20ου αιώνα, υπάρχουν διάφορα είδη συμβασμών. Και μια πολιτική καταπράινσης του Κρεμλίνου ίσως μας οδηγήσει πολύ πιο γρήγορα σε σύραξη από ό,τι φαντάζονται πολύ πολιτικοί ηθήνοντες και κομφορμιστές πολιτικοί άνδρες της Ευρώπης. Η Ρώσο-Ουκρανική σύγκρουση δεν είναι μια τοπική σύραξη, αλλά αμφισβητεί όλη την προηγούμενη πολιτική απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς της Ρωσίας. Και οι συνέπειες αυτής της κρίσης δημιουργούν εστίες ε, πιθανής ε, σύγκρουσης ε, στην Ευρώπη που αυτή τη στιγμή περιορίζονται στην Ουκρανία και έχουν ένα τοπικό χαρακτήρα αλλά τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι δεν θα επεκταθούν και είναι πολύ πιθανό η κατάσταση να εκτραπεί, να πάρει πολύ μεγαλύτερες ζεστές και να έρθουμε σε ανοιχτή αντιπαράθεση Ρωσίας και Δύσης. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Και γύρω από το καθεστώς του Κρεμλίνου βρίσκουμε όλο και περισσότερους που έχουν στοιχηματίσει στην παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανικανότητά της να αντιμετωπίσει την παρούσα οικονομική κρίση. Το Κρεμλίνο περιμένει μια έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια αποτυχία της ζώνης Σέγγεν ή η κατάρρευση του ενιαίου νομίσματος προκειμένου να επιστρέψουμε σε ένα διαμελισμό της ζωνης σεγγεν η καταρρευση του ενιαιου νομισματος προκειμενου να επιστρεψουμε σε ενα διαμελισμο της ευρωπης με βάση ε, τις, ε, τους τέσσερις άξονες Βορρά, Νότο, Ανατολής και Δύσης. Και θέλω να επανέλθουν στη γραμμή ε, νέης όντερ και όχι στην διαφορά Ανατολής Δύσης. Τα γεράκια του Κρεμλίνου δεν περιμένουν με σταυρωμένα χέρια μια κρίση στην Ευρώπη, είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στην δημιουργία προϋποθέσεων για το ξέσπασμα μιας τέτοιας κρίσης. Εξαιτίας λοιπόν της πολιτικής αυτών των γερακιών, η πολιτική της Ρωσίας θα υποδαβλίζει μια κρίση. Διαπιστώνουμε ότι αναγεννιούνται οι παλιές τροτσκιστικές ιδέες για τη μόνιμη επανάσταση με μια νέα τάση και ένα πιο ακροδεξιό και εθνικιστικό χρώμα. Και όλο και μεγαλύτερη λαϊκή υποστήριξη, προκειμένου να συσπηρωθούν όλες οι αναχρονιστικές και εθνικιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό που θέλει ο Πούτιν είναι να κάνει ένα μεγάλο ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας την προπαγάνδα και τη διαφθορά του. Μερικοί θέλουν να μετατρέψουν το σύνθημα «Η Κρυμαία είναι δικιά μας» στο σύνθημα «Η Ευρώπη είναι δικιά μας». Και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρώπη να κινητοποιηθεί, γιατί η ΔΕΜΗ μας περιμένει ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Η σύγκρουση αυτή δεν είναι μια σύγκριση που προκαλείται από τα συμφέροντα της ε, Ρωσίας, αλλά από την επιθυμία ορισμένων να ε, κερδίσουν και να κρατήσουν την εξουσία. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να μείνουμε σταθεροί στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Και αν υπάρχει μία ελπίδα για να αποφύγουμε την κρίση, και την περαιτέρω σύγκρουση, αυτή υπάρχει στην ρωσική γραφειοκρατία που είναι διαυγής, ορθολογική και μη πολιτική. Πρόκειται για ανθρώπους που ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές ε, ε, αξίες και αρχές, αλλά υποχρεούνται να υποταχθούν σε μια διεφθαρμένη και εγκληματική μειονότητα που έχει μονοπολίσει την εξουσία. Η πλειοψηφία της ρωσικής ελίτ αντιλαμβάνεται ότι η παρούσα πολιτική του Κρεμλίνου οδηγεί τη χώρα στον όλεθρο. Βέβαια, έχουν επίγνωση ότι καλό θα ήταν να μην αφήσουν τη Ρωσία να τραβήξει στο χείλος του γκρεμού συμπαρασύροντας και τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά θα πρέπει ο υπόλοιπος κόσμος να στηρίξει αυτή τη λογική φωνή ε, που υπάρχει στη Ρωσία. Γιατί αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, απολυταρχικό καθεστώς, χωρίς ουσιαστικά νόμιμες προπτικές αλλαγής του καθεστώτος. Οπότε στόχος της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν είναι να κερδίσει την εξουσία, γιατί αυτός ο στόχος προς το παρόν είναι ουτοπικός. Στόχος της αντιπολίτευσης είναι απλώς να αντισταθεί στις ε, αντιδραστικές ε, δυνάμεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Κρεμλίνο. Και μάλιστα η συσπήρωση αυτή της αντιπολίτευσης θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες εσωτερικούς και εξωτερικούς. Αυτή τη στιγμή η ρωσική αντιπολίτευση δίνει μάχη όχι μόνο για τη δική της επιβίωση αλλά και για την επιβίωση ολόκληρης της Ευρώπης. Και γι' αυτό η ρωσική αντιπολίτευση χρήζει της ε, υποστήριξής μας. Τι μπορεί να περιμένει ο γνήσιος Ρώσος πατριώτης που είναι ενάντιος ε, στο δόγμα του Πούτιν για την Ευρώπη. Ο πατριώτης αυτός θέλει μία ευφυή, έντιμη και διαφανή πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν λέω ευφυή πολιτική, εννοώ πιο ρεαλιστική πολιτική. Η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι ο Πούτιν δεν ταυτίζεται με τη Ρωσία. Ο Πούτιν κάποια στιγμή θα φύγει. Η Ρωσία όμως θα παραμείνει και θα πρέπει να βρει τη θέση της σε μια ευρύτερη Ευρώπη. Εμείς μετά την πτώση του Βερολίνου αφήσαμε να αναδειχθεί αυτό το φαινόμενο του Πούτιν. Τώρα θα πρέπει να διαχωρίσουμε τον Πούτιν από τη Ρωσία. Άλλο Ευρώπη και Ρωσία, άλλο Ευρώπη και Πούτιν. Και όταν λέω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική εκτός από ευφυής θα πρέπει να είναι και έντιμη, εννοώ ότι δεν θα πρέπει να ε, υιοθετήσει μια απλοϊκή ερμηνεία για τη Ρωσία. Μια καρικατούρα δηλαδή ουσιαστικά της Ρωσίας, ούτε μια μανιχαϊστική ερμηνεία. Δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα, γιατί μερικές φορές φαίνεται ότι και απέναντι στη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μια πολιτική διπλών μέτρων και σταθμών. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι και αυτές ευφύς και έντιμες. Αγαπητοί φίλοι, Έχω πολλούς φίλους στη Ρωσία που είναι πολέμοι του Πούτι και μου είπα να μην ταχθώ κατά των κυρώσεων γιατί κατά τη γνώμη τους αυτές οι κυρώσεις εμποδίζουν το Κρεμλίνο να δείξει ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα, να δείξει ακόμη περισσότερους μυς. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να εφαρμοστούν οι κυρώσεις στη Ρωσία ως χώρα. Καλύτερα να επικεντρώσει τις κυρώσεις στην ρωσική οικονομία. Γιατί αν ο ρωσικός λαός η λογική ότι αν επιδεινωθεί η θέση του ρωσικού λαού θα δει το φως του και θα καταλάβει ποιοι τον κυβερνούν είναι εσφαλμένη. Μια τέτοια πολιτική είναι αμφίβολη αποτελεσματικότητας και θα έλεγα ότι και από στρατηγική άποψη θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικέ συνέπειες. Δεν είναι σκόπιμο ούτε χρήσιμο να απομακρύνουμε το ρωσικό λαό από την Ευρώπη ή να τον κάνουμε να αισθάνεται δυσφορία απέναντι στην Ευρώπη. Θέλουμε οι κυρώσεις να είναι πιο εστιασμένες να στοχεύουν σε συγκεκριμένες οικονομικού οικονομικούς κλάδους, σε συγκεκριμένες προσωπικότητες για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, τρία θέματα πρακτικά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πέραν των κυρώσεων δεν θα πρέπει να διακοπούν οι πολιτιστικές και επιστημονικές ανταλλαγές με τη Ρωσία, γιατί αυτές θα είναι χρήσιμες για τις επερχόμενες γενναίες γιατί να μειώσετε τις πολιτιστικές και επιστημονικές ε, ή εκπαιδευτικές ανταλλαγές με τη Ρωσία. Θα ήταν λάθος. Θα πρέπει να διαφυλαχθούν αυτοί οι πολιτιστικοί και πολιτισμικοί δεσμοί της Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και μάλιστα θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτούς τους δεσμούς για να στρέψουμε τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Μόνο έτσι θα επικρατήσουν οι, οι ευρωπαϊκές αξίες και στη Ρωσία. Θα πρέπει επίσης ε, να γλιτώσουμε τη δίωξη της ρωσικής αντιπολίτευσης από ρωσικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Γιατί ενώ εμείς συζητούμε κυρώσεις κατά του Πούτιν, ο Πούτιν υποδέχεται στο, Κρεμλίνο τον ε, αρχηγό της Ίντερπολ που τον ευχαριστεί για τη συνεργασία του. Επίσης, ε, κάποιοι, κάποια μέλη του διεφθαρμένου καθεστώτος έχουν σχέσεις ε, με ε, Ευρωπαίους ακτιβιστές για να τους αποδείξουν την ορθότητα της θέσης τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα λόγο και δεν μπορεί καν να κρίνει τις ε, άδικες αποφάσεις ε, ρωσικών δικαστηρίων. Θα πρέπει να γλιτώσουμε τους ακτιβιστές από τη δίωξη κάποιων διαφθαρμένων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το Κρεμλίνο κλέβει χρήματα από του Ρώσου φορολογούμενου για να χρηματοδοτήσει κάποιε παράνομε δραστηριότητε στην Ευρώπη ει βάρο των ακτιβιστών. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό για την εικόνα τη Ρωσία. Από τη στιγμή που όλα έχουν ένα τίμημα και όλα μπορεί κανεί να τα ξεγοράσει, αξίζει κανεί να συνεχίσει τον αγώνα του. Σίγουρα το καθεστώς του Κρεμλίνου δεν είναι ισόβιο. Να έχει καμία δεκαετία ακόμη το πολύ διάρκεια ζωής. Γι' αυτό θα πρέπει να συνδυάσουμε τις κοινέ μας προσπάθειες για να αποδυναμώσουμε την ισχύ αυτού του καθεστώτος. Από αυτό θα εξαρτηθεί το μέλλον μας και το μέλλον του καθεστώτος μετά τον Πούτιν. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ο πρόεδρος μιλάει εκτός μικροφώνου. Το λόγο έχει κύριος ε, Κάρας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής με τη Ρωσία. Κύριε Κοντορκόφσκι, αγαπητέ Έλμαρ Μπρόκ, Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρο και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το γεγονός ότι διοργάνωσε αυτή τη συζήτηση αποκινούμε την αντιπροσωπεία για τη Ρωσία και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά δεύτερο, κύριε Κοντροκόφσκι, θέλω να σας καλωσορίσω. Όλοι μας ε, είμαστε ευγνώμονες για τη σαφήνεια των απόψεών σας ε, και για το πρότυπο που είστε για μας. Το ερώτημα που έχω να σας υποβάλω είναι το εξής. Ε, κατά καιρού έχει κανείς την εντύπωση στη Ρωσία. Και έτσι παρουσιάζεται εξάλλου και το θέμα ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Πούτιν είναι ένας τρόπος ε, που, το, που οδηγεί στο να αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς στη Σοβιετική Ένωση και επίσης η εσωτερική κριτική στη Σοβιετική Ένωση προς τον Πούτιν για το λόγο αυτό συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Ερωτώ λοιπόν, τη συζήτηση στη Ρωσία για τον τρόπο συμπεριφοράς και αντίδρασης του Πούτιν και της κυβέρνησης, πώς τον κρίνεται και πώς κρίνεται επίσης και την αντιπολίτευση στη Ρωσία. Επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, έτσι ώστε να στηρίξουμε τις ε, δημοκρατικές προσπάθειες πέρα από αυτά που μας είπατε. Έχουμε την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση έχει αποδυναμωθεί και έχει περιοριστεί περιοριστεί επίσης η δημόσια κριτική κατά τους τελευταίους μήνες. Επίσης, μιλήσατε για ανταλλαγή στον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ συμφωνώ. Εχθές ε, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας ε, της Δούμα μας είπε ότι στη Ρωσία υπάρχει όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους ανταλλαγές γιατί λένε ότι δεν θέλουν να έχουν κανένας είδους επαφή και ανταλλαγή με ένα ε, μόρφωμα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι δικές μου προσπάθειες για ενίσχυση αυτών των ανταλλαγών ε, προσέκρουσαν στον τοίχο των κυρώσεων. Και τρίτον, βεβαίως στο ερώτημα της ε, σύζευξης ρωσικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων Εκεί δεν σας κατάλαβα ακριβώς, δεν κατάλαβα ακριβώς την κριτική σας. Γιατί μιλήσατε έτσι λίγο προσωποποιημένα, δεν το γενικεύσατε. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε λιγάκι πώς ακριβώς σκέφτεστε μία περαιτέρω διαφοροποίηση. Και το τελευταίο με ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πώς ακριβώς την κρίνετε και πώς κρίνεται το λόγο του Memorial κυρίως σε σχέση με την δικαστική διαδικασία και τι έχετε να προτείνετε σε εμά ε, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου στο τέλος του έτους έρεται η απαγόρευση ψήφου για τη Ρωσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Κοντορκόφσκι. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο μας δούλεψε για την ελευθέρωσή σας με ψηφίσματα, με δύο εκθέσεις και μία σύσταση. Ζητήσαμε την απελευθέρωσή σας και χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Οι ερωτήσεις μου μοιάζουν πολύ με τις προηγούμενες, ίσως είναι πιο συγκεκριμένες. Ποια είναι η κατάσταση όσων υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία σήμερα. Έχετε κάποια σχέση εσείς μαζί τους. Μπορείτε να τους βοηθήσετε με το δικό σας κίνημα. Και πώς πιστεύετε ότι αξιολογεί η ρωσική κοινωνία τις δικές μας κυρώσεις, τις κυρώσεις δηλαδή του δυτικού κόσμου. Οι κυρώσεις αυτές πιστεύετε ότι μπορούν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν την κοινή γνώμη στη Ρωσία να μην έχει κακή εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάναμε κάτι διαφορετικό για την κοινή γνώμη πέρα από τις κυρώσεις που αξίζουν κάποιοι αξιωματούχοι της ε, ρωσικής αρχής. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτούς που στηρίζουν τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ κύριε Γκοντορκόφσκι. Για πολλούς από εμά εσείς αποτελείτε σύμβολο για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά της Ρωσίας. Οπότε, συμφωνώ με τις πρώτες ερωτήσεις που ακούστηκαν. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία σήμερα σίγουρα είναι φρικτή. Κάποιες περιπτώσεις θα αναφέρω. Η τάρταρη της Κρυμαίας, για παράδειγμα, το υποκατοχή ε, πρόσφατα έδαφος της Ουκρανίας. Και γνωρίζετε επίσης και την περίπτωση των μητέρων στην ε, Ρωσία. Πώς λοιπόν βλέπετε εσείς τις προοπτικές. Δηλαδή η μάχη έχει ήδη χαθεί, αλλάζει, παίρνει διαφορετική μορφή Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ε, αυτό ήταν ε, καλό παράδειγμα προς μίμηση. Ε, έχουμε 18 ερωτώντες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι. Ο κύριος Λάινεν έχει το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε ο κύριος Λάινεν. Δυστυχώς μιλάει εκτός μικροφώνου ο κύριος Λάινεν. Δεν ακούμε δυστυχώς τίποτα. Το μικρόφωνο είναι κλειστό, δυστυχώς δεν ακούμε. Ναι, τώρα ακούγεται. Λοιπόν, για τρίτη φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ξεκάθαρα λόγια σας. Εγώ είμαι Γερμανός και γνωρίζετε ότι η Γερμανία είναι στόχος της ε, προπαγάνδας ε, του Πούτιν. Έχουν καταπληθεί πολλές ε, προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κοινή γνώμης και είπατε παρά την κριτική που ασκείται η Ευρώπη θα πρέπει κάπως να τα βρει με τη Ρωσία. Και το ερώτημά μου είναι πάνω σε τι να συμφωνήσουμε. Εγώ ξεκίνησα την πολιτική μου σταδιοδρομία με το Willy Brandt, ακριβώς διότι τότε στόχος ήταν να υπάρξει κάποια συνεννόηση, κυρίως με τη Ρωσία. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ πάνω σε τι να συμφωνήσουμε με τον κύριο Πούτιν. Και μία ερώτηση, επειδή εγώ είμαι επικεφαλής αντιπροσωπής με την Κίνα, ο συνάδελφος κύριος Κάρας είναι με τη Ρωσία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτόν τον αναπροσανατολισμό της Ρωσίας που απομακρύνεται από την Ευρώπη και στρέφεται προς άλλου προς την Κίνα. Αυτό έχει ουσία ή μήπως και αυτό είναι ένα είδος ε, προπαγάνδας ε, και παροδικής ε, κρίσης. Επίσης τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί κανείς να κινηθεί. Πολύ με εξέπληξε το ότι είσαστε και από το Ζάρλαντ και είσαστε σύντομος λέει ο πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής maken. Ja, excuus. Ο κύριος Δεσμάκερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κοδοκόφσκι που ήρθατε. Κάποιες από τις ερωτήσεις που είχα να κάνω έχουν ήδη υποβληθεί από τους προλαλήσαντες. Τώρα εσείς μας δώσατε να καταλάβουμε ότι η Ρωσία του Πούτιν, έτσι, έτσι την ονομάσατε, όχι η Ρωσία, η Ρωσία του Πούτιν από ένα αυταρχικό κράτος πλησιάζει να γίνει ένα ολοκληρωτικό κράτος. Και εναντίον αυτού του φαινομένου θέλει να δουλέψει αντιπολίτευση. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο πλήση εγκεφάλων στην κοινή γνώμη. Εσείς πώς θέλετε να αλλάξει αυτή η κατάσταση τη στιγμή που δεν μπορείτε να έχετε παρεμβάσει στα μέσα ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο στη Ρωσία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή η κοινή γνώμη να ενημερώνεται καλύτερα, η αντιπολίτευση να φτάσει καλύτερα, να έχει πρόσβαση στην ε, κοινή γνώμη. Και όσον αφορά τις κυρώσεις, είπατε ότι οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να πλήξουν τους πολίτες. Οι σημερινές κυρώσεις πρέπει να πετύχουν. Έχουμε όμως και το θέμα της τιμής του πετρελαίου. Πώς νομίζετε ότι επηρεάζουν οι κυρώσεις λοιπόν αυτές σήμερα τους Ρώσους πολίτες. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη πρέπει να τη συνεχίσει τις κυρώσεις αυτές και νομίζετε ότι μπορεί να το αντέξει αυτό γιατί πλήττουν και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις ευρωπαϊκές με κυβερνητικέ οργανώσεις. Πώς θα βρεθεί η σωστή ισορροπία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κοντροκόφσκι, είσαστε ο μόνος άνθρωπος σήμερα στον κόσμο που έχει περάσει από τα ρωσικά γκούλακ. Και ο Πούτιν σας χρωστάει 10 χρόνια και θα πρέπει να βρει τρόπο να σας αποζημιώσει γι' αυτό. Η Ρωσία έβγαλε τον εαυτό της από τις χώρες που εμπιστευόμαστε, από τις χώρες που μπορούμε να ονομάσουμε χώρες κράτους δικαίου που σέβονται το διεθνές δίκαιο. Είναι κατανοητό. Περιμένουμε από τη δημοκρατική αντιπολίτευση στη Ρωσία να αντισταθεί στην πολιτική του Πούτιν. Η ερώτηση που έφτασε από το Twitter σε εσά τον Οκτώβριο ήταν η εξή. Θα επιστρέψω την Κρυμαία όταν γίνεται πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και εσείς απαντήσατε. Η απάντησή μου είναι όχι. Όχι επιστροφή δηλαδή. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν το πρόβλημα της ε, Κρυμαίας θα κρατήσει δεκαετίες. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τη θέση σας για την Κρυμαία, γιατί εμείς ποτέ δεν θα δεχτούμε την ε, προσάρτηση και την κατοχή της Κρυμαίας από τις ρωσικές δυνάμεις. Η προπαγάνδα του Κρεμλίνου στην Δύση έχει κάποια επιτυχία με την εξή έννοια ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία λένε ότι η στρατηγική της Ρωσίας είναι κατανοητή και αυτή η προπαγάνδα προέκυψε γιατί στη Δύση έγιναν λάθη, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και σε σχέση με τη Συμφωνία Σύνδεσης. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό και η δεύτερη ερώτησή μου. Είπατε ότι στο Ντόμπας υπάρχει μια περιφερειακή σύγκρουση και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον. Μήπως φοβάστε και εσείς ότι θα συνεχιστεί η εισβολή της Ρωσίας στα ανατολικά, στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Κύριε Κοντοκόφσκι, πραγματικά... Ε, αισθάνομαι ανακούφιση και χαρά που σας ε, συναντώ επιτέλους ε, μετά από τόσα χρόνια που επιθυμούσα. Με εντυπωσιάζει που ο κύριος Πούτιν επιστρέφει σε συμπεριφορά Σοβιετικής Ένωσης με την ΚΑΚΕΜΠΕ να κρατάει τα ίνια της εξουσίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αν και το σοβιετικό στρατιωτικό καθεστώς είχε ε, κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, πιστεύετε ότι θα είχαμε ακόμη την ίδια κατάσταση γιατί συνεχίζονται τα εγκλήματα και κανένας δεν παραπέμπεται ως υπέτειος γι' αυτά. Επίσης, μήπως ήταν λάθος ε, που η Σοβιετική νομιμεκλατούρα έμεινε στην εξουσία παρά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, κυρία Γκριγκούλε. Αξιότιμη κύριε Χονταρκόφσκι, Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση στην μητρική σας γλώσσα. Εδώ, δεξιά. Για να μην χαθεί τίποτα από τη διερμηνία. Είμαι από τη Λετωνία και έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Ποια πιστεύετε θα είναι η συμπεριφορά της Ρωσίας απέναντι στις χώρες της Βαλτικής. Γιατί πρόσφατα είχαμε άσκηση πίεσης ε, κατά των ε, δημοκρατιών της Βαλτικής. Και ποιος πιστεύετε θα είναι ο δικός σας ρόλος ε, στο πολιτικό μελλοντικό προσκήνιο της Ρωσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χοντορκόφσκι, ομολογώ ότι ενστερνίζομαι τις περισσότερες απόψεις και αξιολογήσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, για την Κρυμαία. Δεν έχει δοθεί απάντηση ακόμη. Η Ρωσία αναπτύσσει τεράστιες ποσότητες ε, αμυντικού και ε, επιθετικού υλικού, πυράβλους ε, βραχαίους και μεσαίου βεληνικούς, καταδεκτικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και Ισκαντέρ 300 με μέσο βεληνικές για μεταφορά πυράβλων πυρηνικών. Γιατί πιστεύετε ότι ε, ότι η Ρωσία μεταφέρει τόσε τεράστιε ποσότητες πολεμικού υλικού που διαταράσσει την ισορροπία στη Μαύρη Θάλασσα. Επίση, γιατί πιστεύετε ότι η Ρωσία χρηματοδότησε, χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα σε πολλέ χώρε μέλη. Πιστεύετε ότι κάνει τώρα η Ρωσία αυτό που έκανε στο παρελθόν, το καθεστώ του, του, το ναζί, το νατσιστικό καθεστώ με την πέμπτη φάλαγγα. Πώς ερμηνεύεται αυτή την συστηματική και συστημική αντίδραση και στάση της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Mr. Gurek. Gurek. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ. Είστε ίσως ο πρώτος Ρώσος καλεσμένος μας στην καινούργια κοινοβουλευτική θητεία. Και θα ήθελα επί, τη ευκαιρία να σας θέσω μία ερώτηση στο πλαίσιο των τελευταίων πρωτοβουλειών της Ρωσίας στην ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την, ε, σε σχέση με το ψήφισμα που εξυμνεί τον νατσισμό. Πώς ε, σχολιάζετε αυτά τα θέματα και σχέση με το κομμουνισμό και το σοβιετικό παρελθόν και σε ό,τι αφορά την ομοποίηση του Memorial. Ποια είναι η θέση τους ως προς αυτό, ε, προς τη θέση τους για την παραβίαση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών, θρησκευτικών ελευθεριών, παραβίαση δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Δεν χρειάζεται να μας κάνετε εκτενείς διακηρύξεις, απλώς ε, κάποιες συνοπτικές απαντήσεις θα θέλαμε γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν ερωτηθεί ήδη πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά σε σχέση με την οικονομία, νομίζω ότι κάτι ξέρετε από οικονομία. Μπορεί η Ρωσία να αντέξει τις χαμηλές τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, τις κυρώσεις, ίσως νέες κυρώσεις, τη διαφυγή κεφαλαίων. Τι συνέπειες έχουν όλα αυτά στην πολιτική του Πούτιν, γιατί δυστυχώς πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την προσχώρηση, την προσάρτηση συγγνώμη, της ε, Κρυμαίας, ούτε να επιτρέψουμε στον ε, Πούτιν να συνεχίζει. Θα τα καταφέρει με τα οικονομικά του προβλήματα, τι λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ κύριε Κοντορκόφσκι. Όταν ε, σας είδα την τελευταία φορά ήσασταν ε, μέσα σε ένα κλουβί στο δικαστήριο, στην αίθουσα του δικαστηρίου. Εδώ σας βλέπω και σας χαίρομαι πολύ καλύτερα. Έχω δύο ερωτήσεις. Όταν ε, μιλάτε και μιλήσατε για συμβασμό, τι ακριβώς εννοείτε. Και το δεύτερο που σχετίζεται με τον πρώτο η Ρωσία εκτός από την επιθυμία να αναγνωρίσουμε τις ιμπεριαλιστικές της φιλοδοξίες πέρα από αυτό τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε πραγματικά να επικρατήσει μια ισορροπία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κοδοκόφσκι, θέλω και εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Τι ανάλυση κάνετε εσείς για το 85% που φαίνεται να χαίρει στήριξης στην Ρωσία ο κύριος Πούτιν και για την οικονομική κατάσταση. Αυτά δεν είναι θέματα, οικονομική κατάσταση δηλαδή που θα πρέπει να πλήττουν το ποσοστό στήριξης στον ε, Πούτιν. Τώρα για τις σχέσεις Ρωσίας-Κίνας. Εγώ πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα τα ρωσικά συμφέροντα θα πρέπει να φέρουν τη Ρωσία πιο κοντά στα δυτικά συμφέροντα της Ευρώπης και της Αμερικής παρά της Κίνας. Αλλά εσείς πώς βλέπετε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυτή την προσέγγιση της Ρωσίας με την Κίνα. Σε τι συμφέροντα της Ρωσίας ανταποκρίνεται αυτή η προσέγγιση δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Κοτροκόφσκι. Είμαι Λιθουανός, Ευρωβουλευτές και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν επισκεφθήκατε τη Λιθουανία. Όταν είχαμε διώξει σε βάρος ε, ιδιοκτήτη πετραλοκές εταιρείας και σε μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή πιστεύω ότι είσαστε κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά την εθνική πολιτική, πώς γίνεται από το 2008 όταν είδαμε τη Ρωσία να αλλάζει τη στρατιωτική τη στρατηγική και να προσαρτίζει εδάφη όπως το έκανε στην Γεωργία και την Υπεδνηστερία και τώρα την Ουκρανία. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για συνεργασία με την Ευρώπη ακόμα? Τα κύρια επιχειρήματα είναι τα πυρηνικά όπλα. Ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες της Ρωσίας σε προπαγάνδα. Αν μειώσουμε τις κυρώσεις, τότε βοηθάμε τη Ρωσία να έχει περισσότερα χρήματα να διαθέσει στην προπαγάνδα, κάτι το οποίο οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν από πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι οι Ρώσοι πολίτες θα θυμώσουν ακόμα περισσότερο με τον καπιταλισμό αν ζούνε εν μέσω φτώχειας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, έχουμε δίκιο που αφήνουμε την Ουκρανία μόνη της να αγωνιστεί Υπάρχει αρκετή ενότητα στις βαλτικές χώρες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τόσο μεγάλη πρόκληση. Και στην Ευρώπη υπάρχει ενότητα. Όσον αφορά τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή της Νότιας Ευρώπης, υπάρχει τέτοια ενότητα για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κοδοκόφσκι, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ ελεύθερο, όπως και άλλοι. Να, εδώ είμαι και εμείς αγωνιστήκαμε για την ελευθερία σας. Επίσης, χαίρομαι που κάνετε τη διάκριση ανάμεσα στο Κρεμλίνο και το Λό της Ρωσίας. Και εμείς κάνουμε αυτή τη διάκριση και είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό γιατί θέλουμε κράτος δικαίου και δικαιοσύνης, γι' αυτό θέλαμε να εγκριθεί και ο κατάλογος με τις προσωπικότητες ε, της Ρωσίας, τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Δεν θέλουμε να υπάρχουν καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τιμωρήσουμε. Πώς ε, λοιπόν νιώθει τις επιπτώσεις η Ρωσία και πώς θα τις νιώθει αν η Ευρώπη καταφέρει όντως να μιλήσει με μια φωνή. Δεύτερον, θέλω να ξέρω την άποψή σας για την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία, ότι έκλεισε το μεμόριο, ότι διώχτηκαν διάφορες διεθνείς οργανώσεις. Θέλουμε να ξέρουμε τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά. Περιορίστε πραγματικά πολύ ο ρόλος της ε, κοινωνίας των πολιτών και επιβάλλεται ακόμα μεγαλύτερη προπαγάνδα. Σας ευχαριστώ. Eh, Είμαι εκπρόσωπος της ε, Τσεχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας μίλησατε σήμερα για την Ουκρανία και μας και σας διαβεβαιώ ότι εδώ και μήνες παρακολουθούμε με αμύωτο ενδιαφέρον τα επεισόδια και τις εξελίξεις στην πλατεία Μαϊντάν και επίσης τις ηρωικές μάχες στην κοιλάδα του Ντονέσκ, στον Ντομπάσκ και την υπεράσπιση του αεροδρομίου του Ντονέτσκ με κάθε προσπάθεια. Σίγουρα η, η ελίτ και η διανόηση ήταν ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, μοχλός προόδου και κινητήρια δύναμη. Και εσείς μας μιλήσατε για την ελίτ προηγουμένως. Τι ε, προϋποθέσεις θα πρέπει να δημιουργήσουμε ώστε να αποκτήσουν απήχηση τέτοιες, απόψεις, ώστε να είναι και οι απλοί πολίτες ε, κινητήριοι μοχλή τη αλλαγή και να μην περιμένουμε κάτι τέτοιο μόνο από του διανοούμενους και τις ελίτ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοντοκόφσκι, και εγώ χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Και χαιρόμαστε για την αντίδραση της Ολλανδίας. Λοιπόν, θέλω να ξέρω. Είχατε μια ερώτηση και η ερώτηση είναι εμεί πώ θα φτάσουμε στον Πούτιν και πώς θα φτάσουμε στους πολίτες. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση λοιπόν είναι τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες και όχι τον ε, Πούτιν. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Άλλοι επιχειρηματίες λένε ότι πρέπει να έχουμε κυρώσει και άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε. Εσεί τι λέτε, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Ευχαριστώ Θα κάνω Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ε, πόσο πολύ σας θαυμάζουν στην Ευρώπη κύριε Κοντροκόφσκι. Ε, στρέφουμε το βλέμμα σε εσά ε, ως την ελπίδα ε, για το μέλλον, για τη Ρωσία. Και έχω δύο ερωτήσεις να σας υποβάλω. Η πρώτη είναι, εδώ είμαι αν με βλέπετε, όταν θα γίνετε πρόεδρος της Ρωσίας θα αρχίσετε τη διαδικασία από πουτινοποίησης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση της Ρωσίας, γιατί στην Γερμανία αυτή η διαδικασία κάθαρσης οδήγησε στον Νέο Γερμανία μία από τις πλέον διαφανείς ε, χώρες ε, του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει πολύ σε αυτήν. Μετά το 1991, όταν η, Ρωσία δεν ε, απομπολσεβικοποιήθηκε, αυτό ήταν λάθος. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να στηρίξει κανείς την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση δεν είναι σταθερή. Εσείς λοιπόν, τι πιστεύετε σχετικά με αυτή τη δυνατότητα να ε, σταθεροποιηθεί λιγάκι η αντιπολίτευση στη Ρωσία, περισσότερο από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε κύριε Κοντορκόφσκι η Ρωσία είναι ήδη ένας χώρος αντίδρασης των Ισλαμιστών στην περιοχή του Καυκάσου. Εκεί ζουν περίπου 3 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό δικαιολογεί την ύπαρξη αυτού του ειδικού κράτους ασφαλείας που έτσι κι είναι η Ρωσία. Δυστυχώς ε, ο πρόεδρος μιλάει εκτός μικροφώνου και εμεί δεν ακούμε τι λέει. Δεν μιλάει στο μικρόφωνο ο πρόεδρος. Λοιπόν, κλείσαμε τον κατάλογο των μιλητών. Νομίζω ότι το είπα ήδη προηγουμένως. Την επόμενη φορά να το πείτε έγκαιρο ότι θέλετε να μιλήσετε. Τώρα όμως το λόγο έχει ο κ. Κοντοκόφσκι και είναι ήδη 4 η ώρα και δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις. Θα μπορούσαμε για ώρες ακόμα να συζητάμε Όλη τη νύχτα θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ. Αλλά δεν θέλω βέβαια να καταχραστώ της προσοχή σας περισσότερο. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω όλους όσοι πήρατε το λόγο εδώ σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εδώ και χρόνια έχουν στηρίξει εμένα προσωπικά αλλά και τους συναδέρφους μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αποτέλεσαν θύματα του κατασταλτικού ρωσικού συστήματος. Ειλικρινά σας είμαι ευγνώμων και σας διαβεβαιώ ότι η στήριξή σας μέτρησε πολύ και εξακολουθεί να μετράει πολύ για όλους εκείνους που εξακολουθούν να βρίσκονται στις ρωσικές φυλακές και δυστυχώς πολύ λυπάμαι αλλά παραμένουν πολλοί ακόμα στις φυλακές της Ρωσίας. Ρωτήσατε κάτι για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απόλυτα δικαιολογημένη η ερώτησή σας. Ο Πούτιν έχει μια κάπως παραδοσιακή προσέγγιση όταν τα βάζει με την αντιπολίτευση και τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την Δυτική Ευρώπη κλπ. Προσπαθεί να διχάσει. Διέρη και βασίλευε. Όσοι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί του, του στηρίζει. Όσοι αρνούνται συνεργασία μαζί του, διώκονται από αυτόν. Και όταν τα καταφέρνει, τότε έχει κερδίσει. Είναι ο νικητής. Αν η αντιπολίτευση παραμένει ενωμένη, παρά όλους τους πειρασμούς τους οποίους μπαίνει για να συνεργαστεί με τις αρχές, τότε αναγκάζεται οπότε να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Αυτό έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ενοποίηση, έχει να κάνει με τη στάση του απέναντι στην αντιπολίτευση, τη στάση του απέναντι στους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουν εύκολη ζωή βέβαια, εννοείται. Κανείς από εμά δεν θα περάσει καλά ούτε κι εσείς με τον Πούτιν. Έτσι είναι η κατάσταση όμως και με αυτό κάνουμε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να στηρίξουμε το κίνημα των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς Κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα μέσα που έχουμε, που όμως είναι πολύ περιορισμένα. Για τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις που έχουν ανακοινωθεί παρουσιάστηκαν ως κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Ξέρω ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο ψήφισμα. Αλλά η προπαγάνδα του Κρεμλίνου κέρδισε για άλλη μια φορά. Γιατί δεν υπάρχει αντίσταση από την αντιπολίτευση στην προπαγάνδα αυτή. Οι κυρώσεις είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι κατά κάποιο τρόπο στήριξε το καθεστώς ο κόσμος, επειδή παρουσιάστηκαν έτσι τα πράγματα. Πρέπει όμως να τη δράσουμε, όντως. Αν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που αντιπροσωπεύει ο Πούτιν και σε αυτό που είναι η Ρωσία και ο ρωσικός λαός, τότε τότε πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε τα συμφέροντα, να φανεί ότι τα συμφέροντα του ρωσικού λαού με εκείνα του Πούτιν είναι αντιδιαμετρικά αντίθετα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η διαφθορά. Η διαφθορά είναι πραγματική ληστεία στα ταμεία του κράτους. Πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια στην Ουκρανία. Η δημοτικότητα του Πούτιν έπεσε κατεκόρυφα. Και γιατί? Γιατί η διαφθορά γύρω από τον Πούτιν, του περιβάλλοντός του δηλαδή, ήταν κάτι που δεν μπορούσε πια να δεχτεί ο κόσμος. Ο κόσμος είχε βαρεθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή τη συνεχή διαφθορά με όλες αυτές τις δραστηριότητες του περιβάλλοντος του Πούτιν. Για να ανέβει η δημοτικότητα του Πούτιν λοιπόν, σκέφτηκε να δημιουργήσει την Ουκρανική υπόθεση. Το Ουκρανικό ζήτημα. Οι Ρώσοι δεν έχουν τα μέσα, δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση να ξέρουν τι έχει βάλει στη τσέπη του το καθεστώς του Πούτιν και τι περιουσία έχει στη Δύση. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα βρίσκονται εδώ, στη Δύση, στις δικές σας τράπεζες. Από ό,τι φαίνεται τώρα ένα μέρος τους μεταφέρεται προς την Ασία. Παραμένουν όμως μεγάλα χρηματικά ποσά ακόμα εδώ. Αν λοιπόν τις κυρώσεις αυτές, τις εξηγούσε ειδήσει σαν ηθικές κυρώσεις, σαν κυρώσεις σε βάρος εκείνων που κλέβουν την Ρωσία και ότι έτσι προσπαθούν ε, να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει τα πραγματικά προβλήματα και αν μπορούσαμε να δείξουμε που βρίσκονται οι βίλες και τα περιουσιακά στοιχεία όλων ε, αυτών των ανθρώπων ε, που βρίσκονται στο περιβάλλον του ούτε αυτό θα βοηθούσε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνετε εξάλλου. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την κάθαρση. Η Ρωσία είναι βέβαια μια τεράστια χώρα. Αυτού του είδους ιστορίες όπως αυτή που είχαμε στην Γεωργία δεν θα μπορούσε να λάβει χώρα ποτέ εδώ. Βρίσκουμε επικεφαλής του παρελθόντος που εξακολουθούν να μην θέλουν μια άλλη Ρωσία. Ήταν σφάλμα όταν ε, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση το ότι δεν δικάστηκαν κάποιοι άνθρωποι, έστω και ηθικά, που δεν κρίθηκαν ως υπεύθυνοι των εγκλημάτων του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος και στο κάτω-κάτω ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων αυτών. Στην Ρωσία έχω πει ότι πρόκειται για το 10% περίπου της σημερινής νομακλατούρας. Δηλαδή, καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι. Ενώ στον κατάλογο με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται 114 ονόματα μόνο. Στην Ρωσία θα φοβόντουσαν κανονικά οι άνθρωποι την καταγγελία αυτή, αλλά αυτό παραμένει κάτι θεωρητικό μόνο. Είπε ποτέ η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι ότι δεν θέλουμε καμία σχέση με κίνους που κλέβουν το ρωσικό λαό, που λελατούν τον ρωσικό λαό, δεν το έχετε κάνει, θα μπορούσατε. Και θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερα στοιχεία για το που πάνε τα χρήματα που φεύγουν από εδώ και πηγαίνουν στη Ρωσία. Η δίκη του Γιούκος ε, στη Χάγη ε, είχε σαν αποτέλεσμα να πληρωθούν ε, πάρα πολλά δολάρια από τη Ρωσία για να δικαιωθεί. Εκατοντάδες παραδείγματα θα μπορούσα να σας δώσω και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί σιωπάτε για όλα αυτά. Θέλω να απαντήσω τώρα και σε μια δύσκολη ερώτηση που είναι αυτή για την Κρυμαία. Το έχω ήδη πει και μπορώ να το επαναλάβω και εδώ ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας είναι παράνομη. Παρά ό,τι λόγους μπορεί να έχουμε που να μπορούν να εξηγούν το τι έγινε. Πρόκειται όμως για μια παράνομη πράξη. Συγχρόνως, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι ο ρωσικός λαός στην πλειοψηφία του είναι υπέρ της προσάρτησης αυτής της Κρυμαίας. Πώς λοιπόν μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό καθεστώς είναι δυνατόν να δράσει κατά της ε, βούλησης του λαού. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει να πιστεί ο λαός ότι πρέπει να δράσει διαφορετικά, να βρεθεί δηλαδή ένα συμβιβασμό να του προταθεί. Θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε για παράδειγμα να κάνουμε μια ανεξάρτητη οικονομική ζώνη καταρχήν και μετά να αναφερθούμε στην Ευρώπη χωρίς σύνορα. Η Ευρώπη, Οπότε δηλαδή θα μπορούσε να σκεφτεί λύσεις. Θα χρειαζόντουσαν όμως δεκαετίες για να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Και ξέρετε ότι η Κρυμαία προσαρτήθηκε από ένα δικτατορικό καθεστώς. Δεν είναι δυνατόν ένα δημοκρατικό καθεστώς να κάνει τα ίδια. Λυπάμαι αν δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις, αλλά βλέπω εδώ πολύ αυστηρό τον πρόεδρό σας μαζί μου, τον φοβάμαι, γι' αυτό και θα σταματήσω εδώ. muss immer Rolle des Bad Cop spielen. Πάντα πρέπει κάποιος ε, να παίζει το ρόλο του κακού, αλλά ξέρετε ε, έξω από την πόρτα βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργό του Λιβάνου που υποτίθεται θα έπρεπε να είναι εδώ στις 5 ώρα το απόγευμα. Πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Κοντορκόψκη, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι αυτά που μας είπατε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και εγώ Πιστεύω ότι μπορέσατε να δείτε πόσοι από εμά νιώθουν πραγματική συμπάθεια και κατανόηση προς το πρόσωπό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. <laughs> Damen und Herren, wir sind knapp in der Zeit. Darf ich unmittelbar δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως τη συνεδρίασή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε σήμερα κοντά μας τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. Και νομίζω ότι ο Λίβανος είναι μια χώρα η οποία κατά τις ε, τελευταίες δεκαετίες υπέστη τα πάνδυνα, όσο λίγες χώρες. Και θρησκευτικέ διανέξεις, αλλά και κατά κάποιον τρόπο υπέστη και ένα είδος proxy war θα το αποκαλούσα. Δηλαδή ο Λίβανος με 4 εκατομμύρια κατοίκους αναγκάστηκε να δεχτεί πάρα πολλές θυσίες. Όταν επισκέφθηκα το Λίβανο πριν από 9 περίπου μήνες, δεν ήταν εκεί μόνο οι 300.000 περίπου Παλαιστίνοι που ζουν σε καταβλισμούς εδώ και 60 χρόνια αλλά πέραν από αυτούς υπήρχαν και άλλο ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία. Και 1,1 εκατομμύριο πρόσφυγες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια χώρα. Και αν το απολογίσετε και εσείς στις πατρίδες σας, θα δείτε φτάνουμε σε ε, αποτελέσματα που πραγματικά είναι εντυπωσιακά και δείχνουν με σαφήνεια τι είδους βοήθεια χρειάζεται η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Mr. Elmar Brock. Κύριε Έλμαρ Μπρόκ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής, Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την ευκαιρία που μου δίνεται να είμαι παρόν σε μια συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ο τελευταίο σταθμός μιας επιτυχημένης επίσκεψης της Βρυξέλλες όπου αναζωογονήσαμε την μακροχρόνια φιλία και εταιρική σχέση Λιβάνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την παρουσία μου εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που θα είναι νευραλγικός παράγοντας ε, στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ύψιστο επίπεδο δημοκρατικής νομιμοποίησης, ε, στο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τη μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Και άρα είναι και το ιδανικό μέρος για να απευθυνθεί κανείς ε, στην Ευρώπη και στους λαούς της ε, μέσω ημών των αντιπροσώπων αυτών των, Ευρωπαίων πολιτών. Το μήνυμα που θα ήθελα πρώτα να σας διαβιβάσω είναι ένα μήνυμα φιλίας, ένα μήνυμα που στηρίζεται σε πλούσιους ε, πολιτισμικούς, ιστορικούς και γεωγραφικούς δεσμούς και εγκύτητα. Σας μεταφέρω τη φιλία της πατρίδας μου, του Λιβάνου, που είναι από τις παλαιότερες δημοκρατίες στην περιοχή μας. Το δεύτερο μου μήνυμα είναι μια έκκληση και μια κρούση κόδωνος δίνου. γιατί η κατάσταση στην περιοχή μας είναι ανησυχητική. Η βίαιη σύγκρουση στη γειτονική Συρία έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο και στη δική μου πατρίδα το Λίβανο. Ε, ο Λίβανο ε, φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό ε, σύρων προσφύγων με όλα τα συμπαραβαρτούντα και όλες τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές συνέπειες και τα προβλήματα ασφαλείας. Και ενώ ο Λίβανος κράτησε μια πολιτική ανοιχτών συνόρων από το ξέσπασμα της Συριακής κρίσης κρατήσαμε τη φιλοξενία μας και ε, πραγματικά τραβήξαμε αυτή τη φιλοξενία μέχρι τα άκρα. Κάτι που επιβάρυνε υπερβολικά το λαό μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν κατεπηγόντως μέτρα από τη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσουν τη χώρα μου να μετριάσει κάπως ε, τα πολύ σοβαρά αποτελέσματα αυτής της ε, μαζικής ε, εισρωής προσφύγων που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Θα ήθελα ταυτόχρονα να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για όλη την υποστήριξη που παρήχαν μέχρι τώρα. Βέβαια, η κρίση αυτή είναι άνευ προηγουμένου, γι' αυτό και η αντίδρασή μας αυτή θα πρέπει να είναι πρωτοφανής και άνευ προηγουμένου. Εν τω μεταξύ η Λιβανική κυβέρνηση συνεχίζει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της ε, στην αντιμετώπιση της κρίσης και όχι ε, με κοντόφθαλμο τρόπο και ε, με περιοριστικό τρόπο, αλλά με θέσπιση σαφών κριτηρίων εισδοχής, με σεβασμό του διεθνούς δικαίου σε περιπτώσεις μαζικών εισρών. Η τρομοκρατία είναι μια άλλη τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζει η περιοχή και η χώρα μου. Και ενώ οι τρομοκρατικές ομάδες κάνουν κατάχρηση και καταχρώνται το όνομα του Ισλάμ, που είναι μια θρησκεία ειρήνης, ε, μετριοπάθειας και αρμονίας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην πέσουμε στην παγίδα που εσκεμένα δημιούργησαν οι Ισλαμιστές καπηλεύοντα το όνομα του Ισλάμ προκειμένου να δημιουργήσουν διαιρέσει και διχασμούς και χάσματα μεταξύ των θρησκειών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την προσπάθεια των Ισλαμιστών. Από αυτό εξαρτάται η ασφάλειά μας. Γι' αυτό και οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου κάνουν ό,τι βαρούν και με ηρωικό τρόπο και παρά τις περι περιορισμένες τους δυνατότητες δεν φύζονται προσπαθειών. Έχασαν πολύ τη ζωή τους και πλήρωσαν βαρύ τίμημα, για παράδειγμα κατά την προσπάθεια απελευθέρωση 23 στρατιωτών μας μετά από τον αποκεφαλισμό δύο από αυτών και ε, μία τρίτη εκτέλεση ε, εμψυχρό ενός άλλου ε, στρατιώτη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιμετωπίζουν καθημερινά την απειλή εκπαιδευμένων τρομοκρατών που χρησιμοποιούν μη συμβατικές μεθόδους αντιπαράθεσης. Οπότε η επίλυση της πολιτικής κρίσης στην περιοχή είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Και από αυτή την άποψη το παλαιστινιακό πρόβλημα είναι από βρίσκεται στις ρίζες ε, της απογοήτευσης και μετά από πολύχρονη διαπραγμάτευση ακόμη φαίνεται πόρο να απέχουμε από την επίλυση του προβλήματος και οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να στερούνται ε, τους στοιχειώδους ε, και θεμελιώδους δικαιώματός τους για δικό τους κράτος. Οι αραβικές χώρες ε, το 2002 υπέβαλαν ένα πλήρες πακέτο, μια δέσμη μέτρων για μια συνολική σύναψη ειρήνης καλύπτοντας όλες τις πτυχές της σύραξης. Δυστυχώς ε, το Ισραήλ χρησιμοποιεί δίμευση, κατασχέσεις, ε, ε, αφεστερισμό παλαιστινιακών εδαφών και επικισμούς. Βλέπουμε λοιπόν μια πολύ ανησυχητική συμπεριφορά εκ μέρους του Ισραήλ που διαταράσει και την θρησκευτική αρμονία στην όλη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ καλή θέση και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να στυλιτεύσει και να καταγγείλει αυτές τις, αυτά τα λάθη του Ισραήλ και φυσικά να χρησιμοποιήσει οικονομικά και πολιτικά μέτρα για να προωθήσει μια βιώσιμη συνολική λύση που θα στηρίζεται ε, στις νομοθετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Επίσης, ε, κανείς δεν θα πρέπει να μένει στο απειρόβλητο εφόσον παραβιάζει κανόνες του διεθνούς δικαίου. Στο μεταξύ, το, ο Λίβανος δίνει μάχη για να προασπίσει τη σταθερότητα και τη θέση του. Έχουμε μία κυβέρνηση συνασπισμού ευρύτατη που επικεντρώνεται κυρίως στη διαφύλαξη της ασφάλειας και στην ε, ικανοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των συμπολιτών μας. Έχοντας φυσικά κατά νου την κατεπίγουσα ανάγκη της ε, άμεσης εκλογής του Προέδρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών θεσμών. Φυσικά η αναζήτηση του συμβεσμού δεν είναι πάντα εύκολο έργο. Αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από καθέναν. Το τελευταίο μου μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό, είναι ένα μήνυμα ελπίδες. Το λιβανικό μοντέλο μετριοπάθειας, ανεξιδρυσκείας, ανοχής και ειρηνικής συνύπαρξης ε, λειτουργεί αρκετά καλά. Και παρά τις τεράστιες πιέσεις, ε, τις εντάσεις και τις τριβές που αντιμετωπίζουμε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η χώρα μου εξακολουθεί να είναι κόμβος και υπόδειγμα μετριοπάθειας στην περιοχή. Και μάλιστα πρόκειται για ένα μοντέλο που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και προσαρμοστικό και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον. Μου είπαν ότι ήθεστε να γίνεται συζήτηση μετά από τις παρουσιάσεις. Είμαι στη διάθεση λοιπόν για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Πακνό που ε, ομιλεί εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας ΣΡΕΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και θέλω να μιλήσω όχι μόνο εκ μέρους της Επιτροπής αυτή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, αλλά και ως αντιπρόεδρος της διακοινοβουλευτική Αντιπροσωπείας με τι χώρε ΣΡΕΚ. Όπως το είπατε και το είπε και ο κύριος Μπρόκ, υπάρχει τεράστια μεταναστευτική πίεση εξαιτίας των σύρων προσφύγων που αποτελούν 18% σήμερα του λιβανικού πληθυσμού στη Γαλλία, στη χώρα μου, αυτό σήμαινε 12 με 15 εκατομμύρια ανθρώπους να είχαμε υποδεχτεί. Οπότε, εκ μέρου των συναδέρφων εδώ, σας συγχαίρουμε. Συγχαίρουμε τη χώρα σας για την ε, δέσμευσή της αυτή κύριε Πρωθυπουργέ. Τώρα το επιστημιστικό ε, πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών δεν φτάνει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές πιθανότητες αποσταθεροποίησης εξαιτία της κατάστασης των προσφύγων, οπότε εμένα θα μου φαινόταν ανεύθυνη μια τέτοια στάση. Εμείς πάντως πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε έχετε τη βοήθεια που χρειάζεστε για την υποδοχή των προσφύγων. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Συριακή σύραξη έχει βέβαια και πολιτικές επιπτώσεις στο Λίβανο. Το είδαμε. Είδαμε το Εσμπολά που φεύγει από την πρώτη του εντός αγωγικών αποστολή που είναι η αντίσταση στο Ισραήλ για να στηρίξει στρατιωτικά τον ε, Βασάρι Λασάντ είναι ένα νέο επεισόδιο μεταξύ των Σουνιτών και των Σιτών μετά την δολοφονία τη μασκή που είχαμε το 2005. Οι Σουνίτες του Ντάς όμως ε, ε, ανεβαίνοντας κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύετε ότι οι εντάσεις αυτές οι θρησκευτικέ εξαπλώνονται και θα εξαπλωθούν περισσότερο στο μέλλον ε, στο Λίβανο. Θα ήθελα την απόψή σας από αυτό κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, λέει ο Πρέντα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και για τόσα μας είπατε. Αναφερθήκατε στις δυσκολίες που έχει η χώρα σας σε ένα γενικά πολύ ευαίσθητο περιβάλλον. Εγώ θα επικεντρωθώ στην εσωτερική κατάσταση, αυτή με απασχολεί, γιατί και πάλι είσαστε σε μεγάλη πολιτική κρίση. Ο πρόεδρος Λιμνάν εδώ και μήνες ε, τελείωσε τη θητεία του, δεν υπήρξε συμφωνία για την εκλογή νέου Προέδρου και εσείς ο ίδιος δέκα μήνες χρειαστήκατε για να σχηματίσετε κυβέρνηση. Και τώρα, σήμερα, γίνεται συζήτηση για τη δυνατότητα να αλλάξει ο εκλογικό νόμος. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει σύγκρουση. Ε, αν κατάλαβα καλά για το σύστημα, τίθεται το θέμα εκλογή 64 και 68 μελών του Κοινοβουλίου βάσει ενός αναλογικού συστήματος. Οι υπόλοιποι γίνονται αποδεκτοί με ένα πλειοψηφικό σύστημα. Οπότε πιστεύετε ότι σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο, εντάξει ίσως όχι μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου, αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο χρονικό θα υπάρξει συμφωνία ή θα παραταθεί η κρίση και μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, ε, παραδοσιακό καλωσόρισμα στα αραβικά. Το ερώτημα που αφορά σχετικά με τις δυσκολίες του Λιβάνου. Αναφερθήκατε στο θέμα των προσφύγων που προέρχονται από τη Συρία. Όλοι μας ε, γνωρίζουμε τα προβλήματα της Συρίας και του ISIS και ερωτώ τι κάνει η κυβέρνησή σας για να εμποδίσει την Χεσμπολά να επιδεινώσει την κατάσταση στη Συρία και όσον αφορά στο θέμα του ISIS. Πρέπει να σας πω, για μας είναι δύσκολο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να κατανοήσουμε πώς το κοινό αυτό, ο ISIS, έχει καταλάβει όλες αυτές ε, τις εκτάσεις. Ποιος τους στηρίζει τελικά ε, και πόσο πιστεύετε ότι θα κρατήσει αυτή η σύραξη. Μιλήσατε και για την διένεξη, για το θέμα της ε, Παλαιστίνης και εμείς το εξετάζουμε το θέμα αυτό και θέλουμε το πρόβλημα να επιλυθεί. Πιστεύετε ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους θα βοηθούσε ή θα παρεμπόδιζε την διαδικασία ειρήνευσης στην περιοχή. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κύριε Πρωθυπουργέ εκ μέρους της ομάδας μου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ε, η σκέψη μου είναι στη μικρή αυτή χώρα που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει πια ειρήνη. Υπάρχουν πολλά που αποσταθεροποιούν τη χώρα σας σε καθημερινή βάση και τώρα βέβαια υπάρχει αυτός ο πόλεμος μεταξύ Σιητών και Σουνιτών που διεξάγεται στην περιοχή σας. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, αναφέρθηκε στο Euronews ότι οι δικές σας οι δυνάμεις συνέλευαν τη δεύτερη γυναίκα ε, του ε, αρχηγού των ISIS και ποια είναι η σημασία αυτού έχοντας κυρίως κατά νου ότι 20 ομοιροί κρατούνται από το Ισλαμικό κράτος. Και δεύτερον, μήπως μπορείτε να σχολιάσετε τους ισχυρισμούς ε, του προκουρδικού τουρκικού κόμματος ότι η ISIS έχει ξεκινήσει τις επιθέσεις από την τουρκική πλευρά εναντίον του Κομπάινη και μάλιστα και με βοήθεια των τουρκικών δυνάμεων ίσως και ένα αυτοκίνητο να πέρασε από τα σύνορα και να υποβοηθήθηκε και από τους ελεύθερους σκοποστές. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία και το Κατάρ ε, είναι πώς ακριβώς ε, τίθενται σε σχέση με την απειλή του ISIS. Ευχαριστώ. Η διεθνής κοινότητα, αυτό που ονομάζουμε, που ουσιαστικά είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη ως παράρτημα, δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή. Και επειδή δεν υπάρχει αποτελεσματική δράση ή τέλο πάντων ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες, χρειάζονται πολιτικές λύσεις που εγώ δεν τις βλέπω. η Παλαιστίνη και η ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο είναι ένα μηδέν, γιατί συνεχίζονται οι επικισμοί και παραβιάζονται όλες οι συμφωνίες όπως και της Γενέβης. Είναι η, ο πιο μεγάλος επικισμός χρονικά σε όλη την ιστορία του κόσμου. Στη Συρία η αντιπολίτευση γίνεται αντιπολίτευση στους Ισλαμιστές. Ρωτάω λοιπόν, η άνοδος του εξτρεμισμού, του φανατισμού του Ισλάμ στην περιοχή είναι συνέπεια της απελπισίας, της έλλειψης ελπίδας. Εγώ έτσι νομίζω, επειδή ακριβώ δεν υπήρξαν λύσεις στη Βηρητό για την Παλαιστίνη. Τι λέτε εσείς, έπειτα και ο Λίβανος και η Ορδανία είναι δύο θύλακες που απειλούνται από μια καταιγίδα που έρχεται από το Ιράκ και την Συρία με τρομοκρατία στο Σινά και αλλού μέσα από δημοκρατικές κατά τα άλλα δημοκρατίες. Άλλη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει ρητορικές δηλώσεις και δεν κάνει τίποτα, πώς γίνεται αντιληπτή στη χώρα σας. Πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια μετά τις καταστροφές δεν προσφέρει πραγματική πολιτική λύση. Πώς μας βλέπει λοιπόν η περιοχή. Τέλος, τι σενάριο προβλέπετε εσείς ένα σενάριο έκρηξης ή λύσης. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Πρωθυπουργέ. Το 2008 μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στη λεγόμενη συμφωνία της Ντόχα, οι πολιτικές δυνάμεις του Λιβάνου συμφώνησαν στο πρόσωπο του κοινού υποψηφίου του Προέδρου του Λιβάνου. Στις διαπραγματεύσεις αυτές υπήρξε παρουσία και παρεμβάσεις από τον πρώην Εμμύρη του Κατάρ, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, του σημερινού Προέδρου της Τουρκίας κ. Εντοργάν, των σημερινών Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Αλφα Ισάλ, της Συρίας Μουάλεμ, των πρώην Υπουργών Εξωτερικών της Περσίας Μουτάκη και της Γαλλίας Μπερνάρ Κουσνέρ. Η επιλογή ήταν ο Μισελ Σουλεϊμάν, πρόεδρος του Λιβάνου μέχρι τον περασμένο Μάιο. Από τον Μάιο μέχρι σήμερα, και το τέλο του καλοκαιριού, η Βουλή είχε συνεδριάσει για να εκλέξει νέο πρόεδρο πάνω από πέντε φορέ και ίσω μέχρι σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, να είναι δέκα. Πιστεύετε ότι για την εκλογή του Προέδρου της χώρας σας οι προαναφερόμενες χώρες, δυνάμεις και πρόσωπα του 2008 μπορούν να παρεμβαίνουν για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση με ακέφαλο το Λίβανο και αν δεν μπορούν ποιοι δεν πρέπει ή πρέπει να το κάνουν και με τι ανταλλάγματα. Θα μπορούσα να σας κάνω και άλλες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτή η ερώτηση περιέχει πάρα πολλά ερωτήματα και ελπίζω να μας τα διευκρινίσετε, όπως η ανάμειξη της Χεμπολά, της Χεσμολά στη Συριακή κρίση, τον ρόλο του στρατού του Λιβάνου σε αυτήν και το σημαντικότερο οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στην οικονομία της χώρας και στη ζωή των Λιβανέζων. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Ε, είστε σε φίλους εδώ και πραγματικά η χώρα σας και εσείς ε, ε, χρήζεται και αξίζεται αναγνώρισης γιατί προσφέρετε ασφαλές καταφύγιο σε χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες. Έχω μια διπλή ερώτηση. Μιλήσατε για την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 3 δισεκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φυσικά είναι καλό να στέλνουμε χρήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε το τεράστιο αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα αυτής της μαζικής ε, εισρωής προσφύγων στο Λίβανο και τον κίνδυνο που κάτι τέτοιο ενέχει. Όλα είναι ρηλένδετα στην περιοχή και είναι πολύ σωστά αυτά που είπατε και εύστοχα για την Παλαιστίνη και την ειρηνευτική διαδικασία, που ούτε ειρηνευτική είναι ούτε διαδικασία, δυστυχώς. Και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πραγματικά ιστορικό καθήκον να μην εγκαταλείψουμε το λαό της Παλαιστίνης, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, γιατί ε, πολλές από τις ρίζες του κακού προκλήθηκαν από τις δικές μας χώρες. Ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, όπως είπε ο κύριος Καχάν, ποια είναι τα ωφέλη και οι συνέπειες ε, της μιας θετικής αναγνώρισης. Είδαμε την ψήφα στη Σκοτική Βουλή, στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ε, Γαλλία επίσης συζητά το θέμα, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πώς εκτιμάτε εσείς αυτή τη διαδικασία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια όθηση που δημιουργήθηκε για την αναγνώριση. Και τι θα προτείνατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε για να αναζωογονήσουμε μια αποτελματωμένη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ε, συμφωνώ με όλους αυτούς που σας ευχαρίστησαν για το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα σας ε, κατά την παροχή βοήθειας προς τους πρόσφυγες. Αναμφίβολα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη στηρίζοντας ε, και βοηθώντας αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αν το δει κανείς ψυχρά γεωπολιτικά, ο ρόλος σας είναι καθοριστικός, κυρίως ε, θα ήταν τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε και αυτή να διαδραματίσει γεωπολιτικό ρόλο σε αυτή την τόσο σημαντική περιοχή. Κάτω από αυτό το πρίσμα θα ήθελα την ειλικρινή σας άποψη για αυτά που δεν έκανε η Ευρώπη και για αυτά που η Ευρώπη μέσω της κυρίας Μογκερίνη μπορεί να κάνει. Ως Ιταλός ε, θα ήθελα τη γνώμη σας για τη δράση που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή από την UNIPOL, από την ε, Ιταλική, τις Ιταλικές μονάδες. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος που υπάρχει διείσδυσης του ISIS, ο κίνδυνος αυτός να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ξέρετε, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, μια χώρα που είναι λίγο πολύ εγκαταλειμμένη, οι ένοπλες δυνάμεις, ερωτώ, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον ενδεχόμενο μιας τέτοιας απειλής, γιατί μπορεί να προκύψουν ακόμα μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το Λίβανο. Και η Ευρώπη θα πρέπει να προβληματίζεται σχετικά με αυτή την προοπτική. Μπορείτε να μας δώσετε ίσως κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία που να αφορούν στη διείσδυση του Άιζη στη χώρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για τη χώρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης. Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία σας ε, και την ομιλία σας εδώ. Πρόσφατα πραγματοποίησα επίσκεψη στο Λίβανο και διαπίστωσα και ήδη τη δύσκολη κατάσταση, τη δινή θα λέγα κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα σας, που πραγματικά χρήζει και αξίζει τις αμέριστης υποστήριξής μας. Εδώ και καιρό ε, ο Λίβανος είναι ακέφαλος, δεν έχετε πρόεδρο. Έχω μια ερώτηση παρόμοια με τον συναδέλφου Πρέντα. Πιστεύετε ότι θα ήταν ε, ασφαλέστερο για την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών ε, να ληφθεί υπόψη η πολυμορφία, γιατί η πολυμορφία και η διαφορετικότητα είναι πλούτος ταυτόχρονα για μια χώρα και θα πρέπει να συνεπάρχουν αρμονικά διάφορες ε, εθνότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και κύριε Πρωθυπουργέ. Φαίνεται ότι ο Λίβανος ε, με θαυματουργό τρόπο ε, εδραιώνει τη δημοκρατία του βγάζοντας τα εμπόδια από τους προηγούμενους πολέμους. Δεν κυνηγά μόνο τους Σουνίτες η Χεσμολά, έχει και κυβερνητικέ θέσεις, κυβερνητικού στόχους στο Λίβανο. Θα πρέπει να είμαστε μονομερείς. Επίσης, δημιουργείται αποσταθεροποίηση από τη Συρία και ξέρουμε συγκεκριμένες προσπάθειες χρηματοδότησης. Ε, έχετε εντοπίσει τέτοιες αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Συρίας στο Λίβανο και τι γίνεται, ποια είναι η επίδραση των προσφύγων στην ε, Λιβανέζικη οικονομία. Θα ζητήσετε κατά την επίσκεψη σε αυτή μια περαιτέρω βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου για την συνεισφορά του σε αυτή την ε, σκακέρα της Μέσης Ανατολής. Είπατε προηγουμένως ότι ο Λίβανος είναι με μητροπαθή δύναμη στην περιοχή. Συμφωνώ ένα πρότυπο που αυτή τη στιγμή όμως απειλείται ουσιαστικά. Επανειλημμένα αναφέρθηκε ο κίνδυνος του ISIS αλλά δεν πρέπει να περιζόμαστε μόνο σε αυτό. Ε, θέλω να υπενθυμίσω ε, αυτά που υπόθηκαν από την Ανούζρα πριν από ένα μήνα εκ μέρους του Χεσμπολά, του Αλζουλάνη ήταν οι απειλές ε, και αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε πραγματική σύγκρουση στο Λίβανο, ε, κυρίως ε, ανάμεσα στις δυνάμεις Αλνούστρα και την Χεσπολά. Ακριβώς για να υπάρξει κάποια τιμωρία για την ε, παρέμβαση της Χεσμολά στη Συρία. Παρά λοιπόν τη δύσκολη κατάσταση που αναφέραμε προηγουμένως, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ε, προσφύγων που έρχονται από τη, από τη Συρία και προφανώς και οι άλλοι που προέρχονται από την Παλαιστίνη. Ε, αναφερθήκατε στα πολιτικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, Κατά την άποψή σας, η χώρα σας θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει μία κλιμάκωση της έντασης. Ε, ας το, αφήσουμε τον Άζης ανάμεσα στην Αλνούσντρε και τη Χεσμολά. Και επίσης, τι ρόλο μπορεί, μπορεί να παίχνουν τα Ηνωμένα Έθνη που ήδη βρίσκονται στο Λίβανο. Και άλλη ερώτηση, ο Λίβανος τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό που είναι πολύ δύσκολο, στην αναγνώριση της ε, Παλαιστίνης που όπως ευχόμαστε πάρα πολύ θα μπορούσε να αποτελεί μοχλό έτσι ώστε να επανέλθουν ε, οι δύο πλευρές ε, στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων για να επιτύχουν μία λύση διαρκείας. Ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα, επιστρέφοντας από την διάσκεψη για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στη Συρία, πέρασα τα λιβανοσυριακά σύνορα και έχω την εξή ερώτηση. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε ε, το καθεστώς του Ασάντ που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το Συριακό λαό, την Αλνούστρα, το Ίσης ε, να καταπολεμήσει λοιπόν ο Ασάντ όλους αυτούς τους παράγοντες. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το επόμενο θύμα θα είναι ο Λίβανος και το επόμενο το Ισραήλ. I start by expressing... Θα αρχίσω εκφράζοντας την εκτίμησή μου και τις ευχαριστίες μου για τα θερμά σας λόγια. Άκουσα το καθένα σας με προσοχή και ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο πολλές παρεμβάσεις, τόσες πολλές ερωτήσεις. Είναι κάτι που δείχνει δίχως άλλο το ενδιαφέρον σας, το ότι νοιαζόσαστε για το Λίβανο και για τους Λιβανέζους. Οπότε ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις σας μοιάζανε μεταξύ τους, είχαν τον ίδιο στόχο. Ξέρω ότι έχω περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μου και γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω το χρόνο που θα ήθελα και που θα χρειαζόμουν για να απαντήσω στον καθένα σας χωριστά. Θα αναφερθώ πάντως στα πιο σημαντικά σημεία, τα οποία νομίζω απαντούν λίγο πολύ σε όλες σας τις ερωτήσεις. Πρώτον, για την δικιά μας εσωτερική πολιτική κρίση στο Λίβανο. Ναι, έχουμε εσωτερική πολιτική κρίση. Αποτύχαμε μέχρι τώρα να εκλέξουμε νέο πρόεδρο. Πρέπει να παραταθεί η θητεία του Κοινοβουλίου μας και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε με την κυβέρνηση συνασπισμού να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό πάντως που εγώ μπορώ να πω είναι πως ναι, η δημοκρατία στο Λίβανο έχει λειτουργήσει και σε καλούς και σε κακούς καιρούς. Και εξακολουθούμε με τη δημοκρατία να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μερικές φορές και μερικές να μην τα λύσουμε. Όσο όμως υπάρχει δημοκρατία, ελπίζω ότι σύντομα κάποια στιγμή, όπως κάναμε και στο παρελθόν, έτσι και τώρα θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτή την πολιτική κρίση. Το βλέπω. Είμαι εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανάμεσα σε ευρωβουλευτές που καταλαβαίνουν όλοι πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη δημοκρατία. Και ο Λίβανος έχει μακρά δημοκρατική παράδοση στην περιοχή. Όσον αφορά τώρα την ε, Συριακή σύγκρουση και τις επιπτώσεις της στο Λίβανο. Με ρωτήσατε ξανά και ξανά για το θέμα της ανάμειξης των ολιβανικών πολιτικών κομμάτων στην αντιπαράθεση στη Συρία. Θέλω να σας πω ότι όταν σχηματίστηκε η κυβέρνησή μου, συνασπισμού, παρουσιάσαμε ε, η υπουργική δήλωση για την ψήφο εμπιστοσύνη με ένα, με μία μάλλον θέση κυρίως που ήταν ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και η Εσμπολά συμφώνησε. Και ήταν να διακρίνουμε την δικιά μας πολιτική από τόσα συμβαίνουν στη Συρία. Από τη δήλωση αυτή και μετά Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις δηλώσεις και στην πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτήν την ε, πολιτική η οποία απέτυχε σε μερικές περιπτώσεις, ακριβώς σε αυτές που αναφέρατε κι εσείς. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει από το να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τηρούμε την πολιτική αυτή. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη απάντηση, αλλά ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που δεν βοηθάει καθόλου. Έχουμε τώρα στο ISIS. Άκουσα ερωτήσεις γιατί αναπτύχθηκε έτσι το Άσις, ποιες είναι οι ρίζες του. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, ναι, οι ρίζες είναι ότι δεν επιτρέπουμε την μετριοπάθεια να επικρατήσει στην περιοχή, γιατί η μετριοπάθεια είναι το κλειδί για την ειρήνη. Όσο δεν υπάρχει ειρήνη, όλο και μεγαλύτερο εξτρεμισμό θα έχουμε και όλο και περισσότερη τρομοκρατία. Οι τρομοκράτες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να πούνε στον κόσμο ότι αυτή είναι η Σούπερμαν του σημερινού κόσμου και χρησιμοποιούν έξυπνα τα κοινωνικά δίκτυα, τα μέσα για να προωθήσουν την εικόνα τους. Χρειάζεται μια σοβαρή ειρηνευτική λύση στην περιοχή, γιατί μόνο τότε η μετριοπάθεια θα ενισχυθεί και θα σταματήσει ο εξτρεμισμός. Αυτή την έκκληση σας κάνω λοιπόν και νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε ότι χρειάζεται μια λύση για το Παλαιστινιακό. Ναι, για μας οι Σύριοι πρόσφυγες κατέληξαν να είναι ένα πρόβλημα λόγω του αριθμού τους, γιατί πιεζόμαστε πάρα πολύ. Και γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, περισσότερη στήριξη για τις υποδομές μας, για τους θεσμούς μας. Και γι' αυτό πριν από μερικούς μήνες καθορίσαμε και εγκρίναμε μια νέα προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη μας όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά και αυτούς που τους φιλοξενούν γιατί για να μπορέσουμε να αντέξουμε το βάρος τη προσφυγική αυτής κοινότητα πρέπει να ενισχύσουμε και τη δικιά μας την κοινότητα. Και ακριβώς εκεί είναι που με διμερεί προγράμματα με το Λίβανο μπόρεσε να μας βοηθήσει πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με επιτυχία. Κυρίως και με στρατιωτική βοήθεια, δεδομένου ότι προσέφεραν πραγματογνωμοσύνη στο στρατό μας, ο οποίος έβαλε τάξη στη χώρα παρά τις περιφερειακές εντάσεις. Ναι λοιπόν, κάναμε μεγάλα βήματα και τα κάναμε όχι μόνο για να επανέλθει ο νόμος και η τάξη και όχι για να παραμερίσουμε εκείνους που δεν σέβονται τον νόμο, αλλά για να μπορέσουμε και να ερεμίσουμε τις θρησκευτικέ εντάσεις τις οποίες θέλουν να καταχραστούν οι εξτρεμιστές και να τις χρησιμοποιήσουν υπέρ τους. Μπορέσαμε όμως να έχουμε τη στήριξη που μας πρόσφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί ακόμα να μας υποστηρίξει περισσότερο μέσα από την πολιτική γειτονία, ανοίγοντας νέους δρόμους υπέρ της περιοχής. Και πιστεύω ότι η Ευρώπη τη νιώθει αυτή την ευθύνη. Χρειάζεται βέβαια τη στήριξη και του δικού σας, του Κοινοβουλίου, του νομοθετικού σκέλους. Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να κάνετε. Ναι, όντως η συμμετοχή της Ιταλίας μας βοήθησε πολύ τα τελευταία εννέα χρόνια, μετά από το 2006, και μπορέσαμε έτσι να πετύχουμε ειρήνη και σταθερότητα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Λιβάνου, τον Νότιο Λίβανο πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την ανάγκη που υπάρχει για νέο εκλογικό νόμο στο Λίβανο που θα ενισχύσει τη δημοκρατία μας. Θα ενισχύσει την άσκηση της δημοκρατίας. Θα μπορέσουμε να εκλέξουμε νέο πρόεδρο και θα φέρουμε σε πέρας όλα όσα προβλέπει το Σύνταγμά μας για ελευθερία και κυριαρχία της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσω με το εξής. Παρά την πολιτική μας κρίση, παρά την ένταση στην περιοχή, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι το νομισματικό μας σύστημα το τραπεζικό μας σύστημα είναι ιδιαίτερα επιτυχές. Παρά την κατάσταση. Έτσι μπορούν να γίνουν επενδύσεις στο Λίβανο, γιατί η οικονομία μας είναι ιδιαίτερα δυναμική. Και θα το εκτιμούσαμε όλος ιδιαίτερος, αν το λαμβάνατε αυτό υπόψη, και αν οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνεχίζουν με τα προγράμματα που έχουν στο Λίβανο. Σήμερα το πρωί είχα μια επιτυχή συνάντηση με τον πρόεδρο Γιούνκερ. Συνάντησα και την κυρία Μογκαρίνη και οι δύο εξέφρασαν τη στήριξή τους και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. πέρα από τη διμερή βοήθεια, στηρίζω και την περιφερειακή βοήθεια προκειμένου να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό. Τώρα, για ποιο λόγο αναπτύχθηκε ο εξτρεμισμός αυτός και το ISIS, πιστεύω ότι εν μέρη αυτό οφείλεται στην έλλειψη απόφασης που θα έπρεπε να είχε ληφθεί πριν από δύο χρόνια όσον αφορά τις εξελίξεις στην Συρία. Αν αυτό είχε γίνει πριν από δύο χρόνια και είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη Συρία, δεν θα είχαμε φτάσει εκεί που φτάσαμε σήμερα. Διεθνώς όμως πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η κατάσταση ήταν καταδικασμένη να φτάσει εκεί που έφτασε. Και από τις επαφές που έχω με τους διεθνείς ηγέτες, ήμουν στενομένα Έθνη, στη Γενική Συνέλευση εκεί πριν από λίγο καιρό, με εξέπληξε και με εκπλήσει ακόμα όταν θυμάμαι αυτό που άκουσα από τους μεγάλους ηγέτες να με ρωτάνε εμένα τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε στη Συρία, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει στη Συρία. Μα πριν από δύο χρόνια πρέπει να έχει γίνει και δεν έγινε. Και τώρα όλοι νιώθουν χαμένοι και δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε κάτι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πολιτική λύση είναι αναγκαία στην Συρία και μια πολιτική λύση λαμβάνει υπόψη την σημερινή κατάσταση και προσπαθεί να επεξεργαστεί κάτι. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσουμε σε πολιτική λύση. Σίγουρα όμως χρειάζεται πολύ θάρρος και μεγάλο δυναμισμό και μεγάλη επιθετικότητα διεθνώς για να καταφέρουμε να σταματήσουμε την αιματοχυσία, τον εξτρεμισμό και τη σφαγή που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους λοιπόν και πάλι ε, πρέπει να ξεκινήσουμε και ελπίζω να σας δω και στο Λίβανο αν έχετε την ευκαιρία να έρθετε να βρεθούμε εκεί μαζί. Και χαίρομαι που κάποιος από τους συναδέρφους σας ήταν στον Λίβανο πριν από λίγο καιρό είδε την κατάσταση εκεί. Είδε ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Θα επωφεληθείτε από το χρόνο σας στο Λίβανο και θα μπορέσετε και από πρώτο χέρι να δείτε πώς έχει η κατάσταση εκεί. Είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Και άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Prime ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχόμαστε και σε εσάς και στο λαό σας καλή τύχη και σίγουρα η ISIS είναι ένας παράγων με τον οποίο κανένας δεν θέλει να διαπραγματευτεί. Δεν θέλουμε κανένα συμβασμό. Είμαστε αδιάλακτοι και αμήλικτοι απέναντι στο Ισλαμικό κράτος. Κάτι που κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη γιατί πριν ε, δημιουργηθεί πρόσφατα έδαφο για πολιτικό συμβασμό, πρέπει να γίνουν πρώτα κάποιε στρατιωτικέ ενέργειε. Αυτά σα ευχαριστούμε και καλή σα τύχη. Συνεχίζουμε με το δεύτερο θέμα, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπερναρδίνο Λεόν, που είναι εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω κύριε Λεόν με τη νέα σας ιδιότητα, στο νέο σας αξίωμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προθυμία σας για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στη Νότια Μεσόγειο και η επιδείνωση τη κατάσταση στη Λιβύη ανησυχεί τα μάλα όλους τους ευρωβουλευτές. Και μετά την τελευταία συνεδρίαση τη 17 η Νοεμβρίου του, Υπουργείου, του Υπουργικού Συμβουλίου Εξωτερικών υπευλήθησαν προτάσεις που θα πρέπει να εγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στηρίχθηκαν οι προσπάθειές σας για ενίσχυση του, του εθνικού διαλόγου σε μια περίπλοκη κατάσταση, ειδικά με την ε, απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Λιβύης για την εκλογική διαδικασία. Και μάλιστα σε μια διακήρυξη της 26ης υπήρχε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο του Πρόεδρου τονίστηκε ότι δεν ε, νοείται στρατιωτική λύση στην ε, τωρινή κατάσταση. Θα πρέπει να γίνει διάλογος. Θα σας δώσω το λόγο για μια σύντομη εισαγωγική ομιλία, γύρω στο δεκάλεπτο, για την τρέχουσα κατάσταση στην Λιβύη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεθεί πολιτική διέξοδος από την κρίση. Κύριε Λεόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την επιστροφή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τρία χρόνια που ήμουν μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Πραγματικά αισθανόμουν νοσταλγία για τις Βρυξέλλες. Μπορεί μερικοί ιδιαίτερα συμπατριώτες μου ή από άνθρωποι που κατάγονται από πιο ηλιόλουστες περιοχές ίσως ε, παραξενεύονται που λέω ότι επιθύμησα τις Βρυξέλλες και αισθάνομαι νοσταλγία, αλλά πραγματικά αυτό νιώθω και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων. Όπως ξέρετε η κατάσταση στη Λιβύη είναι περίπλοκη. Και βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τους τελευταίους τέσσερις με πέντε μήνες ε, όταν τον Ιούλιο ξεκίνησαν ε, αντιπαραθέσεις στην περιοχή της Τρίπολης από παραστρατητικές ε, Ισλαμιστικές ομάδες, από Ισλαμιστές αντάρτες ε, που ζήτησαν έξοδο από το αεροδρόμιο της Τρίπολης και είχαμε και τους αντάρτες του Σιντάν και με μια ρητορική αποκλεισμού κάποιων πολιτικών δυνάμεων ε, και ταυτόχρονα μία απόπειρα ε, πολιτικών που βρισκόταν κοντά στο κατάφυλλα να κτίσουν ε, την, τον έλεγχο στη Λιβύη και να παρεκτραπεί η μετάβαση, οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Είχαμε δύο μήνες συγκρούσεων στην Τρίπολη. Ακολούθησε μία περίοδος σχετικής ηρεμίας αλλά ξανάρχισαν οι αντιπαραθέσεις ε, και στη Βενγάζη και σε ανατολικές περιοχές της Τρίπολης, στα όρη της Ναφούζα και αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, η στρατιωτική κατάσταση. Έχουμε ένοπλη σύραξη επιτόπου. Η διεθνή κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένα Έθνη αντέδρασαν σε αυτές τις αντιπαραθέσεις, σε αυτές τις συγκρούσεις και σε αυτή την αστάθεια που δημιουργήθηκε στη Λιβύη και που προβληματίζει ιδιαίτερα την παγκόσμια κοινότητα εξαιτία των τεράστιων συνεπειών και του μεγάλου αντικτύπου που έχει για την Ευρώπη και για τις γειτονικές χώρες. Η αστάθεια της Λιβύης επηρεάζει τις γειτονικές της χώρες. Επηρεάζει την ασφάλεια. Αλλά έχει σχέση με την τρομοκρατία, τη μετανάστευση, τις ενεργειακές ροές. Η Λιβύη βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου. Βρίσκεται στο κέντρο του Νότου. Οπότε οτιδήποτε επηρεάζει τη Λιβύη επιδρά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου επηρεάζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά εγείρει ανησυχίες σοβαρότατες σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε ε, τον πολιτικό διάλογο στο προσκήνιο, να περισσώσουμε την πολιτική διαδικασία και να ανακτήσουμε τη μετάβαση κατά κάποιο τρόπο ε, γιατί όλοι οι πολιτικοί όροι στη Λιβύη έχουν διαφορετική σημασία από τις άλλες γειτονικέ ε, χώρες στην Τινησία μπορούμε να μιλήσουμε για μετάβαση προς τη δημοκρατία. Στη Λιβύη, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο μετάβαση, εννοούμε μετάβαση από μια κατάσταση αναρχίας, ε, έλλειψης κράτους, από την κατάσταση μιας δικτατορίας που κατέστρεψε τους κρατικούς θεσμούς και κατέστρεψε οποιοδήποτε στοιχείο ανοικοδόμησης, πολιτικής ανοικοδόμησης, αλλά κατέστρεψε και την οτροπία, την πολιτική κουλτούρα, την πολιτική παιδεία των Είχε ολέθρια αποτελέσματα το καθεστώς του Καντάφη και αυτά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ακόμη και σήμερα και μάλιστα είναι μερικές από τις ρίζες του σημερινού κακού. Οπότε επαναφορά στη μετάβαση, επαναφορά στην πολιτική διαδικασία, αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η διεθνής κοινότητα. Σε μια πρώτη φάση, σε ένα πρώτο στάδιο, συνεργαζόμαστε με τα μέλη της ε, εκλεγμένης Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι η μόνη εκλεγμένη συνέλευση ε, που έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Ε, εκεί είχαμε μέλη της Βουλής που από την πρώτη στιγμή παρακολούθησαν τη συνεδριάση της Βουλής και έχουμε και μέλη της Βουλής από τη Μισράτα, από την Τρίπολη, από, το, από τη Δυτική Λιβύη, που μποϊκότεραν τις ε, κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις. Αλλά η διαδικασία αυτή διεκόπη όταν στις αρχές του Νοεμβρίου εξέδωσε απόφαση το ανώτατο δικαστήριο της Λιβύης σε μία αμφίσιμη απόφαση δικαστική που δεν δημιουργούσε μια καθαρή εικόνα του θεσμικού χάρτη της Λιβύης. Και μάλιστα οι πολιτικές δυνάμεις και το πρώην Γενικό Εθνικό Κογκρέσο της Τρίπολης έλαβε αυτή την απόφαση ως επιβεβαίωση ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι πια η Λιβική Βουλή και ότι ε, η νομοθετική αρμοδιότητα ανήκει σε αυτό το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο της Τρίπολης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν περιπλάκει όλη η πολιτική διαδικασία. Και όποια και αν είναι η ερμηνεία αυτή τη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και είναι δύσκολο να κάνουμε τέτοια ερμηνεία, για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορούμε αν θέλετε αργότερα στη συζήτηση να τους αναλύσουμε. Πάντως όποια και είναι η ερμηνεία αυτή της απόφασης του Ανωτάτου Λιβικού Δικαστηρίου, η αλήθεια είναι ότι σηματοδότησε μία αλλαγή επιτόπου η απόφαση αυτή. Γιατί καμία από τις δύο βουλές δεν έχει πια αντιπολίτευση, οπότε αν μία από τις αρχές ε, στο διάλογο με τη Λιβύη ήταν η νομιμοποίηση να δημιουργηθεί από τη συμπερίληψη της αντιπολίτευσης, να μην έχουμε δηλαδή δύο ξεχωριστές βουλές, γιατί καμία δεν θα χαίρει της πλήρους νομιμοποίησης, και επιπλέον η αυτοαντίληψη των διαφόρων παραγόντων έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, το Εθνικό Κογκρέσο έχει πολύ ισχυρή, ισχυρότερη σήμερα αυτοαντίληψη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή η διαφορά, αυτή η αλλαγή μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τον τρόπο δράσης μας στη Λιβύη. Επίσης, κάποιοι από τους πρωταγωνιστές του διαλόγου του Γαδαμές 1 ε, με βουλευτές που μποϊκότεραν τη συνεδριάση του Κοινοβουλίου στο, στο Τομπρούκ αφισβήτησαν την απόφαση. Αν και η διεθνή κοινότητα, επειδή ακριβώ είναι αφήσιμο το κείμενο τη δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να επισέλθει στην ουσία αλλά παρόλα αυτά η διεθνή κοινότητα άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει την όλη διαδικασία και τις τελευταίες τρεις εβδομάδες με αυτό το θέμα ασχοληθήκαμε. Τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναγγελθεί μια επαναφορά στην πολιτική διαδικασία. Ευελπιστούμε ότι αυτή η αναγγελία θα γίνει σύντομα. Πολύ πιθανόν τις επόμενες μέρες. Οπότε ή δυνατόν την επόμενη κιόλας εβδομάδα θα επιστρέψουμε στο Καδαμές ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Λιβύης που θα συμφωνηθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη για να συνεχίσουμε την πολιτική διαδικασία. Συμφωνία επί της αρχής υπάρχει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα πρέπει όμως να τελειοποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για να επιβεβαιωθεί αυτή η θέση. Αύριο θα γίνει σε υπουργικό επίπεδο μια πολύ σημαντική συνάντηση στις Βρυξέλλες για να δοθεί υποστήριξη εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας ε, στους πιο σημαντικούς παράγοντες ε, αυτής της ε, επιθυμίας επαναφοράς της πολιτικής διαδικασίας. Οπότε, επανέρχομαι στην αρχική ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι από τη σκοπιά των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά και σε πολιτικό επίπεδο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος της Λιβύης. Σε αντίθεση με άλλες γειτονικές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εταίρος που θεωρείται ουδέτερος στη Λιβύη. Οπότε έχει τεράστια επιρροή και μεγάλη ικανότητα διείσδυσης και στο Τομπρούκ και στην Τρίπολη και στη Μισράτα. Οπότε από πολιτική άποψη είναι σημαντικός συνομιλητής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ειδικοί επεσταλμένοι των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται και συντονίζουν συνεχώς το έργο τους με το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έργο των ΗΠΑ έχουν δείξει πόσο σημαντική είναι η επιρροή τους και πόσο θετική στην πολιτική διαδικασία και από οικονομική άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικότερος εταίρος της Λιβύης. Και μάλιστα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εμπορικών συναλλαγών σε όλους τους τομείς. Αν και όπως ξέρετε, στο επίκεντρο βρίσκονται ενεργειακά προϊόντα. Οι περισσότερε εμπορικέ συναλλαγέ ενεργειακών προϊόντων τη Λιβύη γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριο εμπορικό εταίρο τη Λιβύη. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όχι μόνο την ευθύνη αλλά και την ανάγκη να εξηγήσει στους ε, Λίβιους συνομιλητές τη ότι μόνο με μία πολιτική συμφωνία και μόνο με μία κατάσταση που θα γίνει δεκτή από όλου, θα είναι κοινώ αποδεκτή, θα μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι οικονομικές ροές και αυτές οι εμπορικές συναλλαγές. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση του χάους σε σχέση με το ποιο είναι ο συνομιλητής και η ασάφεια και η αβεβαιότητα με το ποιο ελέγχει τι, τι συμβαίνει με την κεντρική τράπεζα, τι συμβαίνει με την, Ευρω... με Αρχή Επενδύσεων, τι γίνεται με τους αντάρτες και τις παραστρατικές ομάδες που θέλουν να ελέγξουν ε, το πετρέλαιο, εργοστάσια, δηληστήρια, τι γίνεται με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Μερικές ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν μια κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο, αλλά η κατάσταση και η εσωτερική νομική τάξη της Λιβύης αναγνωρίζει το άλλο κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν συνεργασία με λιβικές επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν θέμα όχι μόνο ευθύνη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ανάγκη, αναγκαιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εξηγήσει προ του συνομιλητέ της τη Λιβύη ότι θα πρέπει να επιλύσουν αυτή την κατάσταση και να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία για να εξηγιάνουν τι οικονομικέ του σχέσει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο κύριος οικονομικός εταίρος και με τους υπόλοιπους εταίρους. Η Ευρώπη έχει σημαντικό λόγο και για το θέμα της ασφάλειας, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές που ενεπλάκησαν σε μεγάλο βαθμό στην επανάσταση που οδήγησε στην ανατροπή του Καντάφη. Οπότε και η Λιβύη βλέπει την Ευρώπη ως σημαντικό εταίρο σε αυτή την κοινή κατά κάποιο τρόπο επανάσταση και, την, ε, και ο σημαντικό εταίρος στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης μιας νέας Λιβύης. Οπότε το θέμα της ασφάλειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και το θέμα της τρομοκρατίας, γιατί και η Ευρώπη απειλείται από την παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν σημαντική παρουσία στην ανατολική πλευρά, στη Βεγγάζη, στην Τάρνα, αλλά η παρουσία των τρομοκρατικών οργανώσεων δεν περιορίζεται στην ανατολική πλευρά της Λιβύης. Υπάρχει τέτοια παρουσία και στο νότο της Λιβύης. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται και η ζώνη Σαχέλ συμμερίζεται τις ανησυχίες μας ε, για την κατάσταση στην περιοχή και υπάρχουν συνεχείς ροές. Έγινε λόγος για τα στρατόπεδα εκπαίδευσης τζιχαντιστών στη Νότια Λιβύη αλλά και στη Δυτική Λιβύη. Πολύ λιγότερο βέβαια, αλλά στη Σεβράτα και σε άλλες περιοχές έγινε λόγος για παρουσία τζιχαντιστών που μπορεί να κάνουν επιχειρήσεις και στην Τινησία. Οπότε αυτό το θέμα ανησυχεί σοβαρότατα όχι μόνο τη Λιβύη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, την Τινησία, την Αλγερία, γιατί και η σταθερότητα και η ασφάλεια στην Αλγερία μας προβληματίζει. Οπότε είμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός εταίρος πολιτικός, οικονομικός, στον τομέα της ασφάλειας, με μεγάλη εμπλοκή στην πολιτική διαδικασία. Για τον ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικότατος εταίρος και αυτή τη στιγμή ένας Ευρωπαίος είναι επικεφαλής ε, της αποστολής του ΟΗΕ και μάλιστα ένας Ευρωπαίος που ε, εκπροσώπησε τις χώρες ε, του Νότου και αυτό δείχνει πώς αναγνωρίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το σημαντικό ρόλο και την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ε, δική μου η αξία για το ότι συμμετέχω εγώ σε αυτή, την επικεφαλής τη της αποστολής, είναι αναγνώριση του ρόλου και της ε, επιρροής του Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως ουδέτερος ε, εμψυχωτής και διευκολυντής αναζητά αποκλειστικά και μόνο την πολιτική πρόοδο και τη σταθερότητα στις χώρες του Νότου και αν προκειμένου στη Λιβύη. Οπότε αυτή η τιμή δεν είναι προσωπική, αλλά είναι μια αναγνώριση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σημαντική αυτή η ευκαιρία που δίνεται στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Αν δεν καταφέρει ο λαό τη να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία που θα δημιουργηθεί τις επόμενες μέρες αυτή τη νέα διαδικασία του Γαδαμές 2, αν χαθεί αυτή η ευκαιρία για ανέβρεση πολιτικής λύσης, αν οξυνθούν οι αντιπαραθέσεις, οι συγκρούσεις και η ανασφάλεια, θα πρέπει να μειωθούν, θα μειωθούν οι πολιτικές επιλογές των διαφόρων παραγόντων και θα δοθεί πρωταγωνιστικός ρόλος σε αυτούς ε, που χρησιμοποιούν ε, την στρατιωτική δράση και επέμβαση για την διέξοδο από την κρίση. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν για να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα από τη διεθνή κοινότητα προς τη Λιβύη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει την ευκαιρία να διαμηνήσει αυτή την θέση προς τους λίβιου συνομιλητές ώστε να εμπλακούν με ζέση στην αναζήτηση πολιτικής λύσης γιατί αυτή κατά τη γνώμη μας είναι η μόνη λύση και μάλιστα μια λύση που εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον της Λιβύης αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας και ξεπερνά κατά πολύ τα επιμέρους ατομικά συμφέροντα. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία. Αναφίβολα θα έχουμε στη συνέχεια στη συζήτηση την δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε επιμέρους στοιχεία και να βρούμε τρόπους δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά ο καθένας τώρα για ερωτήσεις και παρατηρήσεις παρακαλώ. Ο κύριος Μιγιά μου έχει το πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Λέον. Ξέρετε ότι είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος. Ο εσωτερικό διάλογο ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και ότι οι αποφάσει του δικαστηρίου οι πρόσφατε έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το διάλογο. Με απασχολεί εμένα το εξή πρώτα απ' όλα. Πέρα από τη δυσκολία του διαλόγου στο εσωτερικό, ούτε και σε διεθνέ επίπεδο φαίνεται να είναι εύκολη η συνεννόηση με τι γειτονικέ χώρε. Είπατε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η βοήθεια από τι γειτονικέ χώρε. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχουν θέσεις που να βρίσκονται κοντά τον ΜΕΝ με τον ΔΕ στην περιοχή με τις γειτονικέ χώρες. 17 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη ακριβώς αυτή η προσπάθεια έγινε να υπάρξει προσέγγιση των θέσεων στην περιοχή. Σε τι βαθμό πιστεύετε εσείς λοιπόν ότι υπάρχει τέτοια προσέγγιση. Δεύτερο, ας μας πείτε για την αυριανή υπουργική διάσκεψη. Περισσότερα το ψήφισμα 2164 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι αποτελέσματα φέρνει τέσσερις μήνες μετά την έγκρισή του. Μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερες χώρες συνεργάζονται. Τι πρώτα αποτελέσματα μπορείτε να πείτε εσείς ότι έχετε εντοπίσει τέσσερις μήνες μετά την έγκριση του ψηφίσματος αυτού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, πρέπει να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Θα μειώσουμε το χρόνο αν βλέπουμε ότι δεν προλαβαίνουμε. Ο κύριος Πανσέτη έχει τώρα το λόγο. Καλώς ορίσατε, Μπερναντίνο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι Δίβοι πρέπει να δράξουν αυτή την τελευταία ευκαιρία και οι Ευρωπαίοι οφείλουν να κατανοήσουν τον όλετρο που προκάλεσαν στη Λιβύη. Γιατί αν δεν το κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι, είναι δύσκολο να το καταλάβουν και οι Λίβοι. Γι' αυτό λοιπόν, ίσως ε, νομίζω θα πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις απλές ευχές. Εχθές είπα ύπατη εκπρόσωπος που ήρθε και μίλησε εδώ στην αίθουσα είπε όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που μπορούν να λάβουν ε, ορισμένες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει υποτίθεται ένα κοινό πλαίσιο. Νομίζω ότι σωστά λέγονται αυτά. Βεβαίως ε, κάποια λάθη τα κάναμε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι καταρχήν έφυγε κάποια χώρα και αν δεν καταλάβουμε αυτά τα λάθη δεν θα καταλάβουμε κατ' ουσίαν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Γιατί υπήρξε η επέμβαση στη Λιβύη και μετά κανείς δεν ασχολήθηκε με τίποτα. Και έχουμε λοιπόν τα λάθη γεωπολιτικά, ενεργειακά, μεταναστευτικά και αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά σχετικά με το χαλιφάτο του Ίζης και την τρομοκρατία. Σωστά όλα αυτά, αλλά τι θα γίνει. Σε επίπεδο αρχής ε, τα εμπλεκόμενα μέρη είπαν ότι θέλουν να συναντηθούν. Αλλά ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης. Βλέποντας την κατάσταση στη Λιβύη, προφανώς και εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες από αυτού και η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εναλλακτική λύση, σχέδιο Β. Δηλαδή, ας πούμε ότι η διεθνής ε, κοινότητα ε, έχει αποφασίσει να παραμείνει στη Λιβύη για να θεωρεί, εφόσον θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι η Λιβύη είναι μια καταστροφή. Το ΝΑΤΟ παρενέβη ε, με τις καλύτερες προθέσεις για να ανατρέψει ε, την φρικτή δικτατορία του Καντάφη. Η Αλγερία είχε μάλλον δίκιο ότι υπάρχει τώρα ο κίνδυνος διαίρεσης της χώρας. Έχω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν, μήπως μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον ισχυρισμό ότι ορισμένα κράτη και το δικό μου έχουν ε, τις βέλτιστες ε, προθέσεις, αλλά κατ' ουσίαν πέρα από αυτό εκπαίδευσαν παραστρατιωτικούς και πολύ εξ αυτών γύρισαν στη Λιβύη και έγιναν Ισλαμιστές και τζιχαντιστές. Απόλυτη δηλαδή αποτυχία. Δεύτερη ερώτησή μου. Όσον αφορά το ρόλο του Κατάρ στη χρηματοδότηση των Ισλαμιστών ε, και των άλλων τζιχαντιστών. Μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει με αυτό. Και επίσης τι συμβαίνει με τον Χαλίφα Χαφτάρ. Ε, δεν ακούσαμε πάρα πολλά για τον δικό του πόλεμο κατά της Συρίας. Και τέλος ε, αναφερθήκατε στην απόφαση των Νότου Δικαστηρίου στην Τρίπολη. Οι δικές μου επαφέ λένε ότι οι ε, δικαστές του Νότου Δικαστηρίου εκφοβίζονται, άρα δηλαδή οι αποφάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν αμερόληπτες. Και κατόπιν τούτου κανείς ε, δεν δεσμεύεται από τη μία αναγνώριση του Κοινοβουλίου του Τομπρούκ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Παρακαλώ. Ο κύριος η Λιβύη για μένα είναι μια χώρα θαυμάσια. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο που βρίσκεται στην Τρίπολη και ουσιαστικά την προσωπεύει το 18% γιατί με τους ψήφους εγκρίθηκε. Ποιος είναι ο συνομιλητής. Είναι αυτός αν δεν είναι πραγματικός ο συνομιλητής, αποτελεσματικός, που έχει τη δύναμη του στρατού κτλ, τότε μιλάμε, κάνουμε μια συζήτηση μεταφυσική χωρίς να μπορούμε να έχουμε καμιά απόφαση επιτόπου. Γιατί αυτό που υπάρχει επιτόπου είναι οι οικογένειες, οι φυλές, οι παραστρατιωτικοί που τελικά ελέγχουν τον πλούτο και όχι μόνο στο βορρά αλλά και στο νότο, το γνωρίζετε καλά. Εσείς βέβαια και βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε εξαιτίας της προσωπικής σας αξίας και αυτό θέλω να αναγνωριστεί. Δεν είναι ατύχημα, το αξίζετε. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω και να σας εκφράσω είναι τη βαθιά μου ανησυχία. Γιατί κάθε τόσο έχουμε και περισσότερες ομάδες που διαπιστώνουμε ότι αυτές κρατάνε τη σχέση με τον πληθυσμό. Πέρα από την ψηφοφορία, μα δεν υπάρχει ψήφος, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν φυλές ε, στην Λιβύη που κυριαρχούν. Εδώ και μήνες λοιπόν εκφράζω την ανησυχία μου και το ξέρετε για τον νότιο τμήμα της ε, Λιβύης που εξάγει όπλα προς κάθε κατεύθυνση και το έχω διαπιστώσει και εγώ και το λέω και το ξαναλέω χωρίς να μου δίνει κανένα σημασία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι βοήθεια αποτελεσματική μπορείτε να προτείνετε αμέσως για να προστατεύσουμε τα σύνορα της Λιβύης με το Τσάντ, τον Ήγυρο. Εντάξει, με την Αίγυπτο γίνεται καλή δουλειά. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη. Αν δεν βοηθήσουμε τον Ήγυρο, το Τσάντ, τον Σουδάν, τότε θα έχουμε τη μεγαλύτερη υπεραγορά όπλων από ποτέ. Η Σοφία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Λόν για την ενημέρωση που μας κάνατε. Στο δελτίο τύπου του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ στι 26 του 2014, μετά την επίσκεψη τη αντιπροσωπεία του στη Λιβύη, το Συμβούλιο Ασφαλεία εξέφρασε τη στήριξή του στον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κύριο Μπερνάντι Νολιού. Καλέσατε τι αντιμαχόμενε πλευρέ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει, καταγγείλατε την αύξηση τη βία, εκφράσατε την ανησυχία σας για την καταστροφή των υποδομών της χώρας, καταγγείλατε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις απειλές κατά των κοινωνικών και πολιτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων των εργαζομένων στον ΟΗΕ, Επίσης καταγγείλατε την παρεμπόδιση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, υπενθυμίσατε την απόφασή σας 2174 του 2014 που ετοιμάζεται να επιβάλλει μέτρα εναντίον αυτών που απειλούν την ειρήνη, την σταθερότητα και την ασφάλεια. Η ερώτηση είναι, μπορείτε να μας πείτε επιτέλους ποιοι είναι αυτοί που εμποδίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λιβύη τόσο καιρό. Και δεύτερον, η κυβέρνηση του Εθνικού Συμβουλίου στην Τρίπολη σας κατακρίνει ότι μεροληπτείτε υπέρ της κυβέρνησης του Κοινοβουλίου του Τον Μπρουκ. Τι απαντάτε επ' αυτού και πείτε μας εάν έχετε συναντήσει τον συνταγματάρχη Χαφτάρ και ποια είναι η άποψή σας για αυτόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και κύριε Λεόν για όλα αυτά που μας είπατε. Πράγματι, ομολογουμένως, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το Σεπτέμβρη εγκρίναμε ένα ψήφισμα όπου περιλαμβάνονται πάρα πολλά από τα ευρωπαϊκά αιτήματα και τότε είπαμε ότι σας στηρίζουμε στην αποστολή σας και στα καθήκοντά σας που είναι να διεξάγετε τον εθνικό διάλογο σε πολιτικό επίπεδο με όλους ε, τους ε, παίκτες με επιρροή. Και ερωτώ έχετε επαφή στους παραστρατιωτικούς και τις ομάδες. Έχουμε μια έκθεση της Amnesty International τέλη Οκτωβρίου όπου αναφέρεται ότι ειδικά στα δυτικά της Λιβύης ε, παραστρατιωτικοί και ένοπλες ε, δυνάμεις ε, επιτίθενται σε πολίτες τους οποίους θεωρούν και μπορούν να θεωρηθούν και εγκληματίες πολέμου. Ρωτώ λοιπόν, έχετε επαφές ε, και τα έχετε συζητήσει όλα αυτά. Το δεύτερο είναι το εξής. Ε, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εσάς ε, να διεξαχθεί πολιτικός διάλογος. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση των μεταναστών στη χώρα. Και τι ακριβώς ε, γίνεται με τους μετανάστες όταν περνάνε τα σύνορα της ε, Λιβύης. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς έχετε κάνει στο πλαίσιο των εργασιών σας. Ο συνάδελφος Καστάλντο έχει το λόγο. Αξιότιμα εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας και κυρίως ε, για τη συνεισφορά σας ε, στη σημερινή συζήτηση. Προφανώς ε, και εγώ εύχομαι η διαδικασία καντάσμε 2 να έχει κάποια δυνατότητα να επιτύχει. Το κοινοβούλιο του Ρομπρούκ, το Μπρουκ, εκπροσωπεί μόνο ένα κομμάτι της χώρας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές ρίζες ανάμεσα βορρά και νότου. Κατά την άποψή σας, πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος να υπάρξει μια ε, κατάτμιση της χώρας κατά τους επόμενους μήνες έτυχε να διαβάσω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τις δηλώσεις ε, του Λίβιου ε, πρέσβη στην Ιταλία, ο οποίος επισημαίνει την αναγκαιότητα της επιστροφής του ΝΑΤΟ στη χώρα, αλλά όχι ως ε, ειρηνευτική δύναμη, αλλά για να βομβαρδίσει. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό αποδεικνύει ότι αποτύχαμε στο ρόλο μας να ε, εκπροσωπήσουμε μια εναλλακτική λύση για να υπάρχει η κοινωνία των πολιτών και η δημοκρατία. Ε, μέχρι τώρα απλά έχουμε δει βομβαρδισμούς. Και γι' αυτό τα είπε αυτά που είπε ο πρέσβης. Άρα δηλαδή είναι σαφές ότι λείπει μια σαφή ε, στρατηγική, έλειπε το 11, λείπει και σήμερα. Κατόπιν, ο ρόλος της Τινησίας. Η χώρα αυτή δέχεται χιλιάδες ε, πρόσφυγες ε, που έφυγαν μετά το 11, αλλά η άνοιξη, η αραβική άνοιξη εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει εκεί. Και τι ρόλο μπορεί να παίξει την νησί για την σταθεροποίηση της δημοκρατίας. Γενικότερα η τιμισία σε αυτή τη σκακέρα έτσι ώστε να δρομολογήσει ανακοχή και γιατί όχι και ειρήνη στην περιοχή. Πρέπει να είσαστε σύντομοι γιατί τελειώς. δεν θα προλάβει να μας απαντήσει ο κύριος Λεόν. Ο κύριος Μποργέτσι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θα περιστώ σε ένα επιχείρημα στο θέμα της μετανάστευσης. Όλοι βλέπουν ότι η χαοτική κατάσταση της, ε, Ολυβής, της Λιβύης καθιστά ακόμα πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς τελικά τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές και ποιος τις ελέγχει. Θα ήθελα να μας ε, πείτε τη δική σας άποψη επ' αυτού του θέματος γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό κυρίως επειδή κάποιος ισχυρίστηκε πολύ σωστά ότι ο νότος της ε, Συρίας ε, είναι ε, αποθήκη όπλων και όλη η κατάσταση συνολικά στη χώρα μας απασχολεί, όχι μόνο του Βορρά, απασχολεί κατάσταση και τις όμορες χώρες. Υπάρχει μια μόνιμη μεταναστευτική ροή και θέλω να ρωτήσω ποιος διαχειρίζεται αυτές τις ροές. Μόνο η παραστρατιωτική και ποιος είναι ο ρόλος των τσιχαντιστών σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τη διεθνή ασφάλεια. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τουλάχιστον στη Δύση τελικά δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα για το τι ακριβώς διαδραματίζεται. Ανταυτού εμείς βλέπουμε να έρχονται συνεχώς μετανάστες, βεβαίως και προς την Ευρώπη, αλλά κυρίως προς την Ιταλία. Βλέπουμε άτομα τα οποία περνάνε μέσα από τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν μας ενισχύει η κατάσταση πάρα πολύ και ελπίζω αυτό να είναι κάτι που να το έχουν υπόψη τους όλοι. Ο κύριος Καν έχει το λόγο. Uh, uh, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε κύριε Λεόν που μας παρουσιάσετε τις απόψεις για το θέμα αυτό. Φυσικά όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει σταθερότητα στη Λιβύη. Φυσικά είναι μια κοινωνία με διάφορες φυλές. Πώς α, πιστεύετε ότι οι γειτονικέ χώρες χρησιμοποιούν αυτή την ε, κοινωνική διαστρωμάτωση και τι ε, ενέργειες γίνονται για να αποφευχθεί η χειραγώγηση αυτή τη κατάσταση. Φαίνεται ότι οι πιστοί στον Καντάφη αρχίζουν και ανασυγκροτούνται. Τι κινδύνους βλέπετε από μια τέτοια συσπήρωση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις, ε, τον καταμερισμό των εδαφών ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, τι εδάφια έχει κάθε ομάδα. Μιλήστε για τζιχαντιστέ. Τι, τι είδου τζιχαντιστέ είναι αυτέ, Είναι του ση, του Ισλαμικού κράτου, τη Αλκάιντα ή κάποια άλλη οργάνωση. Η κυρία Γκόμε, ευχαριστούμε. Ε, Καλώ όρισε και πάλι στο Κοινοβούλιο Μπερναρντίνο. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε τη νέα ιδιότητα ω ειδικό απεσταλμένο της, ε, των Ηνωμένων Εθνών. Το έργο σου δεν είναι μόνο δύσκολο, αλλά είναι και επικίνδυνο γιατί πρόσφατα ε, επέζησες από μία απόπειρα ε, και όπως πολύ διπλωματικά είπες, ε, αυτός ο πολιτικός διάλογος είναι η τελευταία ευκαιρία για τη Λιβύη. Ίσως έχουμε, χάσουμε και Εμεί έχουμε χάσει αυτή την τελευταία ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται ότι μερικοί δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο τη αναζωπήρωσης τη βία εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το ΝΑΤΟ έφυγε πολύ πρόωρα ή πολύ νωρί. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήρθε αρκετά έγκαιρα, αρκετά νωρί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα του SSRDDR γιατί ήταν φανερό από την αρχή ότι αν αφήσουμε αυτού του αντάρτες, αυτή την παραστρατητική ομάδα, ομάδα να κάνει ό,τι θέλει, τι αφήσαμε ξέφραγο αμπέλ, ήταν, ήταν αναμενόμενο ότι θα ε, ανανέωνε του δεσμού τη με την τρομοκρατία μιλούμε για τις γειτονικέ χώρες. Ήδη την Ισία υποφέρει τα πάνδυνα. Πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν εισρεύσει κάτι που δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ε, αλλά ακόμη και η Αίγυπτος που δεν ε, ε, επεμβαίνει, στηρίζει την κυβέρνηση του Μπρουκ η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία που δεν είναι άμεση γειτονική χώρα αλλά είναι επίσης γειτονική. Επίσης ε, η Τουρκία και το Κατάρ που στηρίζει τους αντάρτες ε, στη Μιζράτα που είναι αυτοί που έχουν την εξουσία στην Τρίπολη. Ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, είναι δυνατόν η καλύτερη πολιτική λύση να είναι η διέρεση της Λιβύης στα δύο. Και μία άλλη ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα ο αποθανών βασιλιάς να μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο γιατί ενδεχομένω να μπορεί να επηρεάσει τις ε, συμμορίες Απλά ερώτηση κάνω εγώ, εγώ ερώτηση κάνω. Ο η οικογένεια του ποθανόν της προφανώς, με συγχωρείτε. Μήπως σε τελική ανάλυση η ανατροπή του Καντάφη ήταν λάθος. Σας ευχαριστούμε. Ήρθε η σειρά μου. Δεν μιλάω ως πρόεδρος, αλλά ως μέλος της ΓΚΟΕ, NGL. Μερικές φορές κάποιες αλήθειες ενοχλούν. Και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω παρόλο που ενοχλεί την αποτυχία της επέμβασης του ΝΑΤΟ. Και κρίμα που δεν είχαμε δώσει τη δέουσα σημασία στην Αφρικανική Ένωση και στην πρωτοβουλία της Αλγερίας και δεν είχαμε επιλέξει διαφορετική λύση και όχι την πολεμοχάρη. Τώρα έχουμε απώλεια αμάχου πληθυσμού αθώων, μεγάλη ανθρωπιστική κρίση και την Λιβύη στο χείλος του εφηλίου πολέμου και τη μετατροπή της σε ένα άναρχο κράτος. Με βάση πληροφορίες της Γαλλίας, η Λιβύη χρησιμοποιείται ως βάση για εκπαίδευση τσιχαντιστών από την Αίγυπτο και την Τινησία με την υποστήριξη της Τουρκίας και του Κατάρ. Η Αίγυπτος τα σχήρας της λέει ότι δεν συμμετέχει, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι βοβάρδισαν κρυφά αντάρτικες δυνάμεις. Επίση, μια συνέντευξη του Υπουργού της Τινησίας είπε ότι η Λιβύη είναι ορολογιακή βόμβα για την Τινησία και την Αλγερία. Μας απασχολεί λοιπόν η Λιβύη και, αλλά και το λαθρεμπόριο όπλων γιατί ορολογιακή ε, βόμβα είναι και για μας και για την Αλγερία. Ε, τζιπ 4x4, πυρομαχικά, πύραυλοι ΣΑΜ 7, ε, αντιαρματική πύραυλη, ε, πολεμοφόδια, πυραμαχικά, ακόμη και αεροσκάφη. Δύο αεροσκάφη έχουν εξαφανιστεί από τη Λιβύη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θεαματικές ε, επεμβάσεις στην Αλγερία, Αλγερία και την Συρία. Γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Επίσης, ε, γιατί δεν προσφεύγουμε και στην Αφρικανική Ένωση και στον Αραβικό Σύνδεσμο για ε, να βοηθήσουν για τον ε, εθνικό διάλογο και τι γίνεται με τα κοιτάσματα πετρελαίου που βρίσκονται σε χέρια ανταρτών. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο τώρα κύριε Λεόν. Ευχαριστώ. Πολλές εύκολες ερωτήσεις όπως ό,τι έχει να κάνει με τη Λιβύη. Θα προσπαθήσω γρήγορα να απαντήσω όσο γίνεται περισσότερο σε όλες τις ερωτήσεις. Διεθνή συνεννόηση με τις χώρες του κόλπου και με τις γειτονικές χώρες. Είναι πολύ βασικό. Χωρίς τέτοια συνεννόηση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν περιφερειακοί φορείς που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και δεν μιλάμε μόνο για τις γείτονες χώρες, η Αίγυπτος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια, αλλά μιλάμε και για άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο μακριά από το άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον. Τουρκία, Κατάρ, Εμμυράτα, χώρες δηλαδή που επηρεάζουν σαφώς την κατάσταση. Όλες αυτές οι χώρες στηρίζουν σήμερα την πρωτοβουλία. Συνεπώς, η πρόταση αυτή θα υποβληθεί με την στήριξη Όλο το χωρών που ξέρουμε ότι επηρεάζουν τις διάφορες πλευρές και αυτό είναι θετικό. Όσον αφορά τώρα την αυριανή διάσκεψη, είναι μία διάσκεψη της ομάδας Πέτρες και πέντε. Ήτανε και τρεις μέχρι τώρα, γιατί ήταν οι τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα έχουν προσθεθεί η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Μάλτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί συνεδριάζουν αύριο. Παρακολουθούν από κοντά όλες τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και σίγουρα είναι μεγάλη στήριξη και για μας. Δεν αποκλείουμε κανέναν βέβαια, καθ' άλλο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ανοιχτή Στη Μαδρίτη υπήρξε το 5 και 5 συν, στην Νέα Υόρκη υπήρξε πάλι συνάντηση όπου συμμετείχαν και οι χώρες του κόλπου για παράδειγμα και θέλουμε να υπάρξει και μια νέα τέτοια συνάντηση και μπορεί όντως να λάβει χώρα στη Μαδρίτη. Αυτό δηλαδή που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι με διάφορες μορφές τέτοιες συναντήσεις, με διαφορετικές συμμετοχές, ώστε η διεθνής κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών με διάφορους σχηματισμούς. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να αξιολογήσουμε τα συμπεράσματα, μάλλον αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα από το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών πριν από τέσσερις μήνες. Βλέπετε το ψήφισμα αυτό συμπεριλάμβανε τη δυνατότητα κυρώσεων με ειδικό στόχο άτομα ή ομάδες που δεν συνεργάζονται στην ειρηνευτική διαδικασία ή που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Λιβύης. Είναι μια διαδικασία που έχει αρχίσει η Επιτροπή Κυρώσεων στη Νέα Υόρκη υπό την Ρουάντα. Προσπαθεί να δει ποιοι είναι τελικά είτε από τους στρατιωτικούς που συνέχιζαν να απειλούν ένοπλοι σε κάποιες περιοχές της Λιβύης, αλλά και άλλους από πολιτικές ομάδες οι οποίοι αμφισβητούν, περιπλέκουν, κάνουν ό,τι μπορούν τέλος πάντων για να αποφευθεί η ειρηνική λύση. Αυτή είναι ο στόχος. Η δικιά μου η αποστολή βέβαια δεν εμπλέκεται άμεσα, εννοείται ότι συνεργαζόμαστε κάθε φορά που μας ζητάνε πληροφορίες, αλλά δεν συμμετέχουμε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων. Ελπίζω να μπορέσουμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα, να μπορέσουμε έτσι να τα αξιολογήσουμε πλήρως. Όσον αφορά το περιεχόμενο που ρώτησε ο κύριος Πανσέρη της πρωτοβουλίας κάθε μήνα δύο, είναι μια πρωτοβουλία Το Κανταμές 2 λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με πολιτικούς φορείς, οι προσωπικότητες που συμμετέχουν στην νομοθετική εξουσία, αλλά θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι δημοτικών αρχών, που είναι οι άλλες δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές στη Λιβύη και θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών παράλληλα με άλλα τρία σώματα που θα είναι η παραστατιωτική, άλλοι που έχουν ιδιαίτερο βάρος στη Λιβύη όπως έλεγε και ο κύριος Νάρ και τα πολιτικά κόμματα θα συμμετέχουν. Οι επικεφαλείς των φατριών ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στον Νότο. Στις πόλεις είναι πιο πολύ τα πολιτικά κόμματα που έχουν ε, έντονη παρουσία. Πολιτική, ε, παραστρατιωτική, φαντρίες, πολιτικά κόμματα. Όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία, ελπίζουμε, ώστε να καταλήξουμε σε μία λύση. Είναι τελευταία ευκαιρία και για αυτούς και για την Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπε η Άννα πριν από λίγο. Το πρώτο στάδιο, η πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων προσπαθεί να καθορίσει τον χάρτη πορείας, να υπάρξει εθνική κυβέρνηση και η συνταγματική διαδικασία, η οποία τώρα έχει καθυστερήσει, να συνεχιστεί. Βέβαια το Σύνταγμα μπορεί σύντομα να εγκριθεί και να περάσει με δημοψήφισμα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Το δεύτερο στάδιο τώρα, η δεύτερη φάση, εφόσον πετύχει πρώτη, είναι να αντιμετωπίσουμε τα άλλα εκκρεμούντα θεσμικά ζητήματα. Άρα είναι μια διαδικασία όχι συμμετρική, με δύο διαφορετικά επίπεδα η κυβέρνηση, οι αρχές και τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των πολιτών. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο Β, για να μην πω και Γ, όπως το καταμές 2, μετά το καταμές 1, γιατί η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ που σήμερα δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς αν θα πετύχει διαδικασία ή όχι. Υπάρχουν και άνοπλες δυνάμεις. Χρειάζεται μια ερνευτική διασκέψη κανονικά με τον παραδεισιακό τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό αποτελεί μια ευκαιρία. Δεν είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Η αεροπορία τις τελευταίες δέκα μέρες χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα. Γίνονται μάχες, όπως γνωρίζετε, στη Βεγγάζη. Γι' αυτό δεν ξέρουμε αν θα πετύχει. Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε έτσι κι αλλιώς και άλλες εναλλακτικές στην περίπτωση που η πολιτική διαδικασία δεν καταφέρει να λύσει όλα τα ζητήματα για τον κύριο Τάνοκ. Κύριε Τάνοκ, δεν έχω ακριβείς πληροφορίες για την κατάρτιση αυτή στην οποία αναφερθήκατε. Και εγώ τα διάβασα. Το έχω ακούσει και από Βρετανούς συναδέρφους. Για προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με κάποιους οι οποίοι εμπλέχτηκαν από ό,τι φαίνεται σε κάποιες επιθέσεις. Αλλά ειλικρινά συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχω για κόσμο ο οποίος εκπαιδεύτηκε είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε σε άλλες χώρες και ήταν χατιστές. Δεν το ξέρω. Το ίδιο και για το Κατάρ. Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιες αναφορές, αλλά συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχω. Αυτό μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι το Κατάρ στηρίζει ενεργά την πολιτική διαδικασία και την πολιτική λύση. Όλοι οι φορείς που μπορούν να επηρεάσουν τη Λιβύα να γνωρίζουν ότι βρίσκεται στο χείλος του πλήρους χάους η χώρα και δεν θέλουν να γίνει αυτό. Κανείς δεν θέλει να δει αυτό το πλήρες χάος στη Λιβύη και προσπαθούν να το αποφύγουν. Μετά τη δράση στα Ανατολικά, στη Βεγγάζη με τις πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις, μιλάμε για τρομοκρατία. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά. Είναι παραστατιωτική, δεν είναι μέρος των στρατιωτικών δυνάμων της χώρας. Και πιστεύουμε ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία είναι να χρησιμοποιήσουμε τους κρατικούς θεσμούς. Με ερωτηματικό το λέω αυτό. Δεύτερο ερωτηματικό. Ο κύριος Χάφτερ δεν είναι σαφής για τις προθέσεις του. Τον Φεβρουάριο ο κύριος Χάφταρ έθεσε το ζήτημα των δημοκρατικών θεσμών. Δεν είναι σαφές λοιπόν ποιος είναι ο στόχος του. Χρησιμοποιεί αεροπορικές δυνάμεις και άλλα στρατιωτικά μέσα που δεν στοχεύουν τους τρομοκράτες συγκεκριμένα όπως λέει, αλλά και ε, άμαχο πληθυσμό, οι γειτονιές. Δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την τρομοκρατία ή τους τρομοκράτες. Το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο, γιατί ο κόσμος έτσι ενώνεται εναντίον του. Ο κόσμος που δεν θα πρέπει απαραίτητα να ενώνεται από τη στιγμή που βάλαμε την Σαρία στις τρομοκρατικές οργανώσεις, είδαμε τι έγινε. Έτσι λοιπόν, αυτός ένωσε τον κόσμο εναντίον του. Η διεθνής νομιμότητα είναι εκείνη που είναι πιο αποτελεσματική. Άρα εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Αυτό που κάνει ο κύριος Χάφτερ δεν βοηθάει πολύ πάντως. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να δώσει μια ευκαιρία στην πολιτική διαδικασία και να μην αμφισβητεί την μετάβαση και την οικοδόμηση δημοκρατίας στη Λιβύη. Παρόλο που ξέρουμε ότι αυτό θα πάρει χρόνο και ότι έχει τεράστια ζητήματα να λύσει η χώρα παρόλα αυτά θα έπρεπε να δώσει την ευκαιρία αυτή να το δει σαν ευκαιρία και εκείνος. Τέλος, όσον αφορά τις αποφάσεις, όπως έχω ξαναπεί, θα είναι δύσκολο να τοποθετηθούμε για διάφορους λόγους. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι και οι πόνιες για το ότι το δικαστήριο πήρε τις αποφάσεις αυτές με εκφοβισμό, με την πίεση από παραστατητικούς στη Λιβύη, όλα αυτά είναι αλήθεια. Συγχρόνως όμως είναι αλήθεια όλους τους τελευταίους μήνες. Η Λιβύη είχε παραστατητικούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ήταν πάντα μία πρόκληση. Θέλω να πω δεν είναι κάτι καινούριο. Η φύση των παραστατικών αυτών μπορεί να άλλαξε στην Τρίπολη, αλλά υπάρχουν και από άλλες περιοχές και άλλη προέλευση. Δεν είναι εύκολο λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα δεν είναι νομικό, είναι πολιτικό, γιατί ακόμα και αν υπήρχε σαφής ερμηνεία των αποφάσεων του ενότατου δικαστηρίου, πάλι θα υπήρχε πολιτικό ζήτημα στη Λιβύη. Συνεπώς η Λιβύη πολιτική λύση πρέπει να βρει και αυτό πρέπει να ενθαρρύνει και η διεθνής κοινότητα. Έρχομαι Τώρα στην ερώτηση του κυρίου Νάτ, νομίζω ότι απάντησα στην πρώτη, ότι το ΚΑΔΑΜΕΣ s S2 θα έχει παρουσία με τις φατρίες, ε, τις τα κτλ. Τώρα για το δεύτερο είναι μια περίπλοκη ερώτηση. 4.000 χιλιόμετρα έχει σύνορα η χώρα με το Σαχέλ, άρα υπάρχουν και όλες οι προκλήσεις του Σαχέλ. Τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικά κλπ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι χώρες που γνωρίζετε πολύ καλά νοτίως της Λιβύης είναι εύθραυστες, ευάλωτες και έχουν ελάχιστες δυνατότητες να περιορίσουν το λαθρεμπόριο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια έχει μια αποστολή συνόρων η οποία ελπίζω πολύ γρήγορα να μπορέσει να επιστρέψει στη Λιβύη και να συνεισφέρει στον έλεγχο των συνόρων και να είναι αποτελεσματική. Βέβαια είναι μια περιοχή που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε γιατί χώρες αυτές ούτε Λιβύη ούτε οι γείτονε χώρε νοτίως της Λιβύης έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν από μόνες τους αυτές τις προκλήσεις. Ποιοι φταίνε, ποιοι είναι αυτοί που αντιτίθεται στην πολιτική λύση. Έχετε ακραίους, εξτρεμιστές και στα δύο στρατόπεδα. Έχετε στους Ισλαμιστές εκείνους οι οποίοι είναι κοντά στους τσιχατιστές στο ριζοσπαστικό Ισλάμ που δεν στηρίζουν πολιτική λύση. Αυτό είναι σαφές. Και έχουμε δει κάποιους από αυτούς πρόσφατα σε διαδηλώσεις στο, σε εκδηλώσεις μάλλον στο Λίβανο, σε επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Εθνών και άλλα. Είναι βέβαια μια μειοψηφία ευτυχώς. Οι περισσότεροι μετροπαθείς Ισλαμιστές στηρίζουν την πολιτική λύση. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη μεριά, Έχετε επίσης ομάδες μετριοπαθών, που είναι η πλειοψηφία, και στηρίζουν τον πολιτικό διάλογο, αλλά έχετε και μία μειοψηφία εξτρεμιστών που πιστεύουν ότι όλοι οι Ισλαμιστές είναι τρομοκράτες και δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί τους. Προς το παρόν Ιδίως όταν πρόκειται για άνοπλες δυνάμεις και τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία της Λιβύης, παραστρατιωτικούς κτλ. είτε από την άλλη μεριά, δυστυχώς δεν βλέπουμε να στέλνουν κανένα σημειογραφής ότι θα στηρίξουν την πολιτική διαδικασία. Νομίζω ότι έτσι απάντησα και για τις παραστατιωτικές οργανώσεις. Ποιος θα μιλήσει μαζί τους δεν έχει νόημα να προωθήσουμε μία ε, πολιτική συμφωνία αν συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις ή να επιβάλλουν. Δεν είναι δυνατόν από ένοπλη δράση να πετύχεις κάποια συμφωνία. Βέβαια, στην κρίση της Λιβύης δεν μπορείς να δώσεις λύση αν δεν χρησιμοποιήσεις και αυτούς τους ανθρώπους σε ένα βαθμό. Γι' αυτό και λέμε ότι θα συμμετέχουν στην διαδικασία που αρχίσαμε. Για τον κύριο Καστόλτο. Κίνδυνος διχασμού και κατακαιρματισμού. Μα ήδη είναι διχασμένη η Λιβύη. Ήδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο κοινοβούλια, δύο κυβερνήσεις, πλειοψηφία με στρατιωτική επιρροή τη μισή χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, ότι είναι μια ευκαιρία και για τη Λιβύη και για τη διεθνή κοινότητα. Έχει δίκιο η κυρία Γκόμε που λέει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία και για εκείνου και για μας. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Το νότιο τμήμα έχει το δικό του δυναμισμό, το είπε και ο κύριο Νάτ πριν. Ο κίνδυνο, λοιπόν ήδη υπάρχει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό και τους διχασμούς. Αν δεν είναι ενωμένη Λιβύη δεν θα είναι βιώσιμη. Αυτό πιστεύουμε. Συμφωνώ μαζί σας ότι πληρώνουμε το τίμημα της αποσίας της διεθνούς κοινότητας από το 2011 και βέβαια και η Τινησία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο γιατί στα δυτικά και στην Τρίπολη έχει επιρροή. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές, οι μαφίες, νομίζω το κάνουν. Δεν είναι πολιτικές ομάδες ή παραστατιωτικές που πρέπει να κατηγορηθούν για αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Η κατάσταση όμως είναι δύσκολη και δύσκολο να αξιολογηθεί γιατί επικρατεί κλίμα ανασφάλειας, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει διοίκηση. Και πρέπει πρώτα να λυθούν όλα αυτά για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση και σε αυτή την ερώτηση. Ποιες είναι οι μαφίες και πώς στηρίζονται για την εμπορία αυτή ανθρώπων κάπου χίλιοι το χρόνο. Οι τζιχαντιστές παίζουν σημαντικό ρόλο. Απαντάω επίσης και στο ποιοι είναι οι τζιχαντιστές. Οι περισσότεροι τζιχαντιστές στην Λιβύη δεν είναι ομάδες που έχουν εκφράσει ε, κάτι που να δείχνει ότι ανήκουν στο ISIS. Αλλά υπάρχει χούντα κουβενή οι οποίοι έχουν εκφράσει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα μικρό φαινόμενο, μας ανησυχεί βέβαια, αλλά υπάρχουν άλλες ομάδες που δεν έχουν εκφράσει τη σύνδεσή τους με το ISIS, μπορεί να το κάνουν βέβαια η Ελσαρία στην Βεγγάζη και στην Τέρνα έχουν εμφανιστεί και υπάρχουν και άλλες το Ελσας Ισλάμ, οι μάρτυρες του Ιουσαλήμ και άλλες ομάδες που μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτή την κατηγορία. Δεν υπάρχει παρουσία μελών του καθεστώτος του Καντάφη εκτός από κάποιους ίσως στην ε, Τρίπολη και Ισλαμιστές που προέρχονται από τον Κατάφη. Όχι, δεν υπάρχει σημαντική τέτοια δύναμη του παλιού καθεστώτος. Προωθούμε τον πολιτικό διάλογο γιατί είναι ένας πολιτικός διάλογος μεταξύ αυτών που πρέπει να συμμετέχουν στο μέλλον μιας δημοκρατικής Λιβύης. Επιμένω ότι εμεί δεν πιστεύουμε ότι εκπροσωπούνται τέτοιε ομάδε του παλιού καθεστώτο, παρόλο που σα λέω, μεμονωμένα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να παρεύουν και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την ε, σύγκρουση αυτή για να επαναφέρουν το καθεστώς του Καντάφη, αλλά είναι πολύ μακριά. Άννα, νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου. Θα το επαναλάβω ότι χωρίς τη διεθνή στήριξη είναι αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία επιμένω στις χώρες κλειδί στηρίζουν τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ζωτική σημασία ρόλο. Δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που κάναμε και κατά το παρελθόν και που εσύ πολύ σωστά επανέλαβες και μας θύμισες. Δεν υπάρχει λύση αν είναι διχασμένη η Λιβύη, επίσης είναι προφανές για μένα. Οι συγγενείς του βασιλετρίστα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο και ε, επειδή μπορούν να επηρεάσουν κάποιες φατρίες ε, της ε, δύση που μπορούν να αποτελέσουν μέρος της μελλοντική λύσης, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον στη μοναρχία, στη Λιβύη. Δεν το βλέπω. Και έπειτα δεν νομίζω ότι ήταν εσφάλμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπήρχε εναλλακτική να κρατηθεί το καθεστώς του Καντάφη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει γίνει με άλλο τρόπο, καλύτερα ή χειρότερα, αλλά κατά τη δικιά μου την προσωπική γνώμη, η εναλλακτική ήταν τα στατεύματα του Καντάφη που βρισκόντουσαν στην είσοδο της ε, Βαγκάζης ή που θα κάνανε σφαγή στην πόλη ή θα γινόταν αυτή η επίθεση, θα άλλαζε η κατάσταση και οι επαναστάτες, όπως έγινε, θα κέρδιζαν. Κατά την δικιά μου ταπεινή γνώμη, δεν υπήρχε χρόνος για διπλωματική πρωτοβουλία. Μακάρι, μακάρι να υπήρχε, μακάρι να ήταν δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι η διπλωματική οδός δεν είχε χρόνο, για τα στατέματα του Καντάφη ήταν ήδη στις πύλες. Και οι ειδικέ δυνάμεις μάλιστα του Καντάφη ήταν μέσα στην πόλη. Αλλά, πάση περιπτώσει, ποτέ δεν θα το ξέρουμε με σιγουριά. Υπάρχει συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Σήμερα πάω στην Αντίσα Μπέμπα για μια συνεδρίαση που θα γίνει αύριο της ομάδας επαφής με την Αφρικανική Ένωση για τη Λιβύη, με τις χώρες της περιοχής. Αύριο στο Σουδάν επίσης συνεδριάζουν οι γείτονε χώρες για να συνεργαστούν με τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών και για να δούμε τι πρωτοβουλίες έχουν εκείνοι. Τέλος, όσον αφορά την αγορά πετρελαίου και την χρήση των περιουσιακών στοιχείων από το πετρέλαιο, ενεργειακούς φόρους και άλλους. Το συζητήσαμε, θα συζητηθεί αύριο στην Υπουργική Συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα. Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί ιδιαίτερα με τη δυνατότητα χρήσης τέτοιων περιουσιακών στοιχείων από κάποιες ομάδες. Οι οικονομικές συνέπειες είναι βέβαια πολύ σημαντικές για όλους τους διεθνείς φορούς και πρέπει να το αποφύγουμε είναι η δουλειά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεόν. Καλή τύχη, καλή επιτυχία. Γιατί αν επιτύχεις εσύ, η επιτυχία θα έχει αντίκτυπο στη Λιβύη, στο λαό της Λιβύης και σε όλους όσους υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Πρόκειται για την έκθεσή μου, μια τεχνικής φύσεως ε, έκθεση, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος το λόγο επ' αυτού. Από ό,τι βλέπω όχι. Κατόπιν τούτου να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Όχι ακόμα. Δεν ψηφίσατε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια εργασία του. και λύει τις συνεδρίες. Γεια σας. Was? Soll doch mit Durchschlagskraft vorgetragen. Ne?